Αν δούμε τι συμβαίνει αν τον κόσμο, βλέπουμε ότι το 2014 το DRC ε, η λαϊκή δημοκρατία του Κονγκό είχε τεράστιες ε, τεράστια ανάπτυξη ε, που είναι μια όμως πολύ φτωχή χώρα στον κόσμο, από τις πιο φτωχές. Η οικονομική ανάπτυξη όμως δεν σημαίνει ότι όλοι μοιράζονται αυτή την ευημερία ε, ή δεν σημαίνει καλές δημοκρατικές δομές ε, και παρέμεινε η χώρα αυτή φτωχή. Ε, πώς θα φτιάξουμε ένα συνεκτικό όλο είναι ε, το ζήτημα. Χωρίς καλούς θεσμου δεν υπάρχει ε, ανάπτυξη. Λοιπόν, έχουμε διάφορους εμπειρογνώμονε εδώ για να μας βοηθήσουν να δούμε πώς θα το υλοποιήσουμε το SDG. Η Έλλης δεν μπόρεσε να έρθει λόγω οικογενειακών υποχρεώσεων. Εγώ λοιπόν ε, θα, είμαι, θα προεδρεύσω το πρώτο πάνελ. Έχουμε διάφορους ομιλητές από διάφορες οργανώσεις για το πρώτο πάνελ που θα συζητήσουμε το, την εμβέλεια και τη γένεση του SDG 16. Έχουμε τη Σάρα Λίστερα από το UNDP, από το Κέντρο Διακυβέρνησης του Όσλο, είναι διευθύντρια εκεί. Έχουμε την... Ε, η κυρία Λότε Κνούτσεν δεν ήρθε εδώ. Ο, ο κύριος ε, Φιλιμπέρτο Τσεριάνι είναι ε, συντονιστής του ΙΕΣ και έχουμε και, ένα, και τον Ζαν Λουί Βιλ ε, που, είναι, που ασκεί χρέη διευθυντή από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Γενική Διεύθυνση Ντεύκο. Σας ευχαριστώ που ήρθατε εδώ. Ε, θα αφήσω τη Σάρα να εξηγήσει ίδια την, ε, το UNDP, το πρόγραμμα αναπτύξή του ΟΗΕ. Το θέμα είναι τι θα αλλάξει τα επόμενα χρόνια με, τους, ε, με, το στόχο της, με το SDG 16. Η Σάρα είναι η πρώτη και μετά θα δώσω το λόγο στους υπόλοιπους ομιλητές. Σας ευχαριστώ για την πρόσκληση. Είμαι διευθύντρια στο UNDP, στο πρόγραμμα ανάπτυξη του ΟΗΕ και στο κέντρο του Όσλο για την ε, διακυβέρνηση που είναι ένα κέντρο για την παγκόσμια πολιτική, για την εφαρμοσμένη έρευνα και το διάλογο ε, για την ε, διακυβέρνηση σε μεταβατική φάση. Συνεργαζόμαστε με διάφορους συναδέλφους στο UNDP και με άλλους συναδέλφους που ασχολούνται με το, που δουλεύουν στο, στον για τον στόχο 16 και εστιάζουμε στο πώς θα μετρήσουμε το στόχο αυτό. Ε, το θέμα είναι πώς θα εφαρμόσουμε αυτό το στόχο, όπως είπε και η Λίντα. Ε, θα κάνω τρεις, παρα, τρεις παρατηρήσεις. Ε, καταρχάς είναι πώς προέκυψε ο, ο στόχος 16, από πού προέκυψε, γιατί με, έχει σημασία και συνεχεία τι πρόοδο έχουμε σημειώσει προς την εφαρμογή του. Θα προσπαθήσω να απαντήσω και τη δύσκολη ερώτηση που μου έθεσε η Πρόεδρος. Λίγες παρατηρήσεις για τη γένεση του στόχ 16 από που προέκυψε. Πριν μιλήσω για τη διαδικασία διαπραγμάτευσης, και δεν θα μπω σε πολλές λεπτομέρειες, θα ήθελα να κάνω μια μικρή ιστορική αναδρομή. Ο, η δήλωση της χιλιετίας είχε πολύ ισχυρή γλώσσα για τη δημοκρατική διακυβέρνηση, για την ε, συμμετοχική, δημοκρατική διακυβέρνηση, ε, για τα ανθρώπινα δικαιώματα, την ε, ελευθερία ε, από το φόβο της βίας. Θα πρέπει να καταβάλουμε κάθε προσπάθεια, έλεγε, ούτω ώστε να προωθήσουμε την δημοκρατία και το κράτος δικαίου και τα αναγνωρισμένα, διεθνώς αναγνωρισμένα ανθρώπινα δικαιώματα και θεμελιώδεις ελευθερίες. Ισχυρή γλώσσα, αλλά δεν εφαρμόστηκαν αυτά. Δεν υπήρχε στόχος της χιλιετίας για τη διακυβέρνηση, για την ε, δημοκρατία. Γιατί. Δύσκολο να απαντήσουμε για πολλούς λόγους. Ορισμένοι πιστεύουν ότι υπήρξαν πολιτικές αντιστάσεις. Αλλά τα περισσότερα θέματα ήταν, ε, βασικά δεν υπήρχε δυνατότητα μέτρησης ε, πριν από 15 χρόνια. Είναι σημαντικό να το καταλάβουμε αυτό στα πλαίσια της σημερινής συζήτησης για το SDG 16. Παρά το γεγονός λοιπόν ότι δεν υπήρχε ε, MDG, ειδικά για, την, ε, για τα φόρμα δικαιώματα, τη δημοκρατία και τη διακυβέρνηση, διάφορε χώρε αποφάσισαν να δημιουργήσουν τον δικό του ε, MDG, τον δικό του στόχο, τον 9. Η Μογγολία, η Αλβανία, το Λάο και άλλοι ανέπτυξαν το δικό του στόχο, το MDG 9, που αφορούσε τα εθνικά θέματα διακυβέρνηση, ασφάλεια και έθεσαν στόχου, ούτω ώστε εθνικό επίπεδο να του υλοποιήσουν στην περίοδο δημιουργή, ε, υλοποίησης των στόχων της χιλιετίας. Στην περίοδο ανάμεσα στη θέσπιση των αναπτυξιακών στόχων χιλιετίας και τη συζήτηση που έγινε για τους στόχους της βιώσιμης ανάπτυξης, ε, υπήρξαν ορισμένε αλλαγέ που κατέστησαν, ήταν προϋπόθεση για τη δημιουργία του σκοπού. Καταρχάς, αναγνωρίσαμε ότι η έλλειψη ε, ειρήνης ε, με ένταξη και δικαιοσύνη εμπόδιζε τη βιώσιμη ανάπτυξη οι συγκρούσεις, οι πόλεμοι κτλ. έχουν πολλαπλές επιπτώσεις. Το καταλαβαίνουμε αυτό σήμερα. Ε, δεν υπήρχαν ε, αποτελεσματικοί θεσμοί ε, που να λογοδοτούν και να εξασφαλίσουν ε, οικονομική, κοινωνική και περιβαλλοντική πρόοδο. όλα αυτά αναγνωρίζονται στην, σε μια δήλωση, στη δήλωση του Ρίος Plus 20 το 2012. Ε, καθώς και σε άλλες διεθνείς δηλώσεις και αναφορές. Υπάρχει μία αναγνώριση ότι η ανάπτυξη και η ειρήνη πάνε μαζί, χέρι-χέρι και όχι χώρια. Η αρχική διαδικασία διαβούλευσης ε, για την ατζέντα μετά το 2015 ε, παρακολουθούσε την ειρήνη και την ανάπτυξη χώρια. Ε, μετά όμως αναγνωρίστηκε ότι δεν μπορούμε να αντιμετωπίσουμε αυτά τα δύο θέματα χώρια γιατί είναι αλληλένδετα. Και νομίζω ότι γίνεται ακόμα μια ε, συζήτηση στην ε, κοινότητα που ασχολείται με την ανάπτυξη και στον ΟΗΕ για το πώς ε, αντιμετωπίσουμε αποτελεσματικά τους τομείς αυτούς. Επίσης υπήρξε μεγάλη τεχνική πρόοδος και πολλά παραδείγματα από όλο τον κόσμο και στην Αφρική για το πώς μπορείς να μετρήσεις στοιχεία της διακυβέρνησης ε, ότι ήταν εφικτό κάτι τέτοιο, με, να το κάνεις με πολύ αυστηρό και επιστημονικό τρόπο. Αυτά ήταν η προϋπόθεση για να δημιουργηθεί ο στόχος 16. Η διαδικασία διαπραγμάτευσης του στόχου 16 ήταν περίπλοκη και ορισμένες φορές πολύ δύσκολη. Αλλά υπάρχει μια, υπήρξε μια τεράστια κινητοποίηση της κοινωνίας των πολιτών γύρω από αυτό το στόχο που ήταν πολύ σημαντικό αυτό. Και επηρέασε την συμφωνία για το στόχο. Ένα παράδειγμα που ξέρετε πολύ, στην επισκόπηση ο κόσμος μου, μία ειλικρινής ε, κυβέρνηση ε, που να λογοδοτεί, αυτό ήταν ε, ένα πράγμα που θεώρησαν πάρα πολύ σημαντικό εκατομμύρια συμμετεχόντων. Σε πολλές συναντήσεις υψηλού επίπεδου ε, είπαν ότι θα πρέπει να υλοποιήσουμε τις προσδοκίες των αυτών που συμμετείχαν, των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών, των πολιτών κτλ. Λοιπόν, αυτά για να σας πω που προήλθε ο στόχος 16. Πάμε τώρα στο δεύτερο κομμάτι ε, της παρουσίασής μου, γιατί έχει σημασία. Ο στόχος 16, όπως ε, λέμε συχνά στον ΟΗΕ, δεν είναι μόνο ένα πολύτιμο και σημαντικό στοιχείο, μια σημαντική φιλοδοξία, αλλά και ένας ε, βασικός στόχος προϋπόθεση για να τη υπάρξει ατζέντα για τη βιώσιμη ανάπτυξη. Η ατζέντα 2030 λέει ότι δεν μπορεί να υπάρξει βιώσιμη ανάπτυξη χωρίς ε, ειρήνη και, όχι, και δεν μπορεί να υπάρξει ειρήνη χωρίς βιώσιμη ανάπτυξη. Ε, μια κυβέρνηση χωρί αποκλεισμού, που ενσωματώνεται και επικονίζεται στο στόχο 16, είναι προπόθεση για την υλοποίηση όλη τη ατζέντα και σημαίνει ότι πρέπει να γίνουν κοινέ προσπάθειε και συνεργασία μεταξύ κυβερνήσεων, ε, κοινοβουλίων, ε, ΜΜΕ, οργανώσεων κοινωνιών πολιτών και διαφόρων φορέων. Κάτι άλλο σημαντικό για τον στόχο 16 είναι ε, ότι είναι το τμήμα ε, μιας παγκόσμιας ατζέντα που συμφώνησαν τα κράτη και που είναι κτήμα πια της διεθνούς κοινότητας με έναν τρόπο που δεν έχει ξανασυμβεί στο παρελθόν. Στο παρελθόν οι κυβερνήσεις θεωρούσαν η διακυβέρνηση συγγνώμη, ήταν κάτι το οποίο ε, επέβαλε ο ανεπτυγμένος κόσμος στις αναπτυσσόμενες ε, χώρες. Το SDG 16 όμως άλλαξε άρδινα αυτή την ε, λογική και συνειδητοποιούμε τώρα ότι όλες οι χώρες έχουν μια κοινή ευθύνη για το στόχο 16. Ένα σημαντικό στοιχείο του στόχου 16 είναι ότι μας δίνει ένα πλαίσιο εφαρμογής ούτω ώστε να ασχοληθούμε και να δουλέψουν πάνω σε διάφορου άξονε, το ανθρωπιστικό, το αναπτυξιακό, ανθρώπινα δικαιώματα, επίτευξη ειρήνη κτλ. Χάρη στο στόχο λοιπόν, ε, το έχουμε συμφωνήσει αυτό διεθνώς. Επίσης είναι σημαντικό να πούμε ότι υπάρχουν διάφορες αρχές εντός του στόχου που απεικονίζονται στο στόχο, αλλά που δεν αφορούν αποκλειστικά το στόχο 16. Υπάρχουν σε όλη την ατζέντα και όλη η ατζέντα πρέπει να θεωρηθεί ως ε, μία ενιαία και αδιέρετη ατζέντα. Υπάρχουν πολλοί στόχοι της ατζέντα του 2030 που έχουν να κάνουν με τη βία, την δικαιοσύνη, την ε, ένταξη, πράγματος χάρη. Ο στόχος 4.7 ε, μιλάει για την πρόθεση μιας κουλτούρας ειρήνης, ε, χωρίς βία, ε, την παγκόσμια ηθαγένεια και την, την πολιτιστική ποικιλομορφία. Ο στόχος 5.2 5,2 μιλάει για την συμμετοχή των γυναικών και την, τον ηγετικό ρόλο των γυναικών. Ε, ο στόχος ε, 16 μιλάει για την καλή διακυβέρνηση, αλλά ε, πάντως στην ατζέντα υπάρχουν στοιχεία του στόχου 16. Οι στόχοι του Goal 16, του SDG 16, καλύπτει ε, βία, ε, κράτος δικαίου, παράνομη χρηματοδότηση και κυκλοφορία όπλων, διαφθορά, ε, ουσιαστικές ελευθερίες, αντιπροσωπευτική λήψη αποφάσεων κτλ. Τα κοινοβούλια είναι πολύ σημαντικό στοιχείο για την υλοποίηση του G16, γιατί είναι ένας από τους μηχανισμούς για την εξασφάλιση μια διακυβέρνηση χωρί αποκλεισμού. Οι φορεί και τα θεσμικά όργανα που ασκούν έλεγχο έχουν ιδιαίτερη ευθύνη για να εξασφαλίσουν αυτή την ένταξη. Ε, η διαδικασία μέτρηση ε, μα δίνει κάποια αναλυτικά στοιχεία τα οποία είναι σημαντικά να χρησιμοποιηθούν δηλαδή, ούτω ώστε να εφαρμόσουμε πολιτικέ για να βελτιώσουμε τη ζωή των ανθρώπων. Υπάρχουν διάφορε προκλήσει με τη μέτρηση και δυσκολίε με τη μέτρηση του στόχου. Ε, ορισμένοι δείκτε είναι απλοί και υπάρχουν δέσμε δεδομένων που μπορούν να χρησιμοποιηθούν. Κάποιοι δείχτες είναι πάρα πολύ περίπλοκοι γύρω από το στόχο και χρειάζονται μία μεθοδολογία για συλλογή των δεδομένων. Ε, και δεν υπάρχουν αποκλειστικά στοιχεία, αλλά υπάρχει μια διαδικασία στο Διεθνές Στατιστικό Σύστημα για να αντιμετωπίσουμε αυτά τα θέματα. Η δουλειά συνεχίζεται και, συνεχι... και θα μπορούσα να σας δώσω περισσότερα στοιχεία αν χρειαστεί στη συνέχεια της συζήτησης. Αυτό είναι ε, μια απάντηση στο γιατί μετρά, ε, έχει σημασία ο στόχο αυτό. Τέλο, τι πρόοδο έχει σημειωθεί προς την εφαρμογή του, μέχρι στιγμής τουλάχιστον. Υπάρχει μεγάλη δραστηριότητα σε διάφορα επίπεδα, σε διάφορους τομείς, για να υποστηρίξουμε την υλοποίηση του SDG 16. Η εφαρμογή σε εθνικό επίπεδο φυσικά είναι ευθύνη των εθνικών φορέων. Το UNDP ως τμήμα του συστήματος του ΟΗΕ και με παρουσία σε 170 περίπου χώρες ε, δεσμεύεται να υποστηρίξει την εφαρμογή του στόχου και συνεργαζόμαστε με εταίρους σε όλα τα επίπεδα, παγκόσμιο, περιφερειακό, εθνικό, υποεθνικό. Σε επίπεδο χώρας υπάρχουν διάφορες πρωτοβουλίες, πολλές πρωτοβουλίες ε, που προωθούμε, θα σας δώσω λίγα παραδείγματα. Παραδείγματος χάρη σε εταιρική σχέση με την Open Governance, και την Community of Democracies ε, υποστηρίζουμε ε, την παρατήρηση σε διάφορες πιλωτικές χώρες ε, της εφαρμογής του στόχου 16, ούτω ώστε να δούμε πώς μπορούν αυτά να χρησιμοποιηθούν για να προωθηθούν διάφορες πολιτικές. αυτό σημαίνει και την ανάπτυξη ενός εθνικού δελτίου επιδόσεων που βασίζεται σε διάφορους δείκτες από το εθνικό, περιφερειακό και παγκόσμιο επίπεδο. Σε επίπεδο χωρών κάνουμε διάφορες προσπάθειες ούτως ώστε να προωθήσουμε πούμε, τις γυναίκες σε θέσεις κλειδιά ας πούμε, στην Αρμενία ε, θέλουμε να τις προωθήσουμε, προωθήσουμε την εκλογή τους στα δημοτικά συμβούλια. Στην Παπούα Νέα Γουινέα, ε, έχουμε συνεργαστεί με έναν πάροχο τηλεπικοινωνιών, ούτω ώστε να δημιουργηθεί ένα πρότυπο σύστημα αναφορά με SMS ε, που θα στέλνει ειδοποιήσεις, προειδοποιήσει για διαφθορέ σε, ένα κρατικό φορέα επιτήρηση. Ε, Επίση, στην Τινησία ε, υποστηρίζουμε το Υπουργείο Εσωτερικών, ε, ούτω ώστε να υπάρχει ένα νέο μοντέλο ε, στην αστυνομία ε, που θα βασίζεται στην ιδέα της παροχής υπηρεσίας στο δημόσιο. Επίσης, ε, σε υποεθνικό επίπεδο υποστηρίζουμε την τοπική διάσταση των SDG. Ε, καταλαβαίνουμε ότι το SDG 16 μπορεί να εφαρμοστεί μόνο αν ε, συμμετάσχουν και οι τοπικοί φορές, φορείς, όχι στην εφαρμογή μόνο, αλλά και στην παρατήρηση και στην ε, καθώς και στην θέσπιση της, α, της ατζέντας. Στη, στην πράξη αυτό σημαίνει υποστηρίζουμε τοπικούς φορείς, α, του δίνουμε πρακτικά εργαλεία, και γραμμέ κτλ. Σε περιφερειακό επίπεδο υποστηρίζουμε την, τον εμπειρισμό των εμπειριών, ε, τη συγκέντρωση των γνώσεων. Ε, θα συναντηθούμε στην Καρταχένα για να μιλήσουμε για την ε, υλοποίηση του στόχου SDG 16 ε, στην περιοχή αυτή. Επίσης, σε παγκόσμιο επίπεδο, το UNDP συνεργάζεται με άλλες υπηρεσίες του ΟΗΕ, με διάφορους ε, φορείς, ε, σε πολυμερέ, διμερέ επίπεδο, με διάφορες οργανώσεις, κοινωνίες πολιτών, ακαδημαϊκούς και τον, δημόσιο, και τον ιδιωτικό τομέα. Επίσης, υποστηρίζουμε μια παγκόσμια συμμαχία για την αναφορά προόδου, για την προώθηση ειρηνικών δίκαιων ε, κοινωνιών χωρί αποκλεισμού. Είναι ένα δίκτυο ε, με πολλούς φορείς για την υποβολή εκθέσεων για την εφαρμογή του SDG 16. Υπάρχουν τα τεχνικά και μεθοδολογικά στοιχεία για τη μέτρηση των δικτών του SDG 16. Υπάρχουν πάρα πολλά παραδείγματα τα οποία θα μπορούσαμε να συζητήσουμε ε, στην φάση ερωτήσεων απαντήσεων. Τώρα απλώς σας έδωσα μία έτσι, πρόγευση. Έχω φέρει και ένα φυλάδιο, ε, μπορείτε να το πάρετε. Υπάρχει και ένα newsletter που παράγουμε ε, ούτως ώστε να σε ενημερώσουμε για τις δραστηριότητες γύρω από το SDG 16. Σας ευχαριστώ για το χρόνο σας και πιστεύω ότι θα, κάνουμε και άλλα, θα πούμε και άλλα πράγματα στη συζήτηση που θα ακολουθήσει. Ευχαριστώ πολύ. Στην αρχή ξέχασα να πω κάτι. Αρχικά έχουμε και κάποιους ε, καλεσμένους. Από την Μιανμάρ, ε, Βερμανία, ο κύριος Κούντι Μιν. Εργάζεται ε, στο Κοινοβούλιο της Μιανμάρ και μετά Βάιλιν Σο. Σας ε, καλωσορίζουμε εδώ στην σημερινή μας ε, συνεδρίαση. Ευχαριστούμε. Um, and, um, we, it would be good to exchange how, how you και καλό θα είναι να ε, αλλάξουμε, ανταλλάξουμε απόψη σχετικά με την εργασία των ε, κοινοβουλίων μας. Γιατί βλέπουμε ότι ενισχύεται η δημοκρατία στη χώρα σας και αυτό είναι πολύ θετικό. Το δεύτερο που θέλω να πω είναι ότι δεν συμμετέχουν πολλοί ευρωβουλευτέ σήμερα, αλλά έχουμε και άλλου ε, παρευρισκομένου. Αν έχετε εσεί λοιπόν ερωτήσει, μπορούμε να τι ε, δεχθούμε, αρκεί να είστε σύντομοι. Θα ακούσουμε λοιπόν ερωτήσει και από άλλου, αν υπάρχουν ε, καυτά ερωτήματα. Αυτά λοιπόν για το ιστορικό του ε, στόχου 16. Τώρα θα δώσουμε το λόγο στον κύριο Τσεριάννη Σεβρικόντι. Ή κύριε Φιλιμπέρτο πιο απλά. Για την απάντηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τι θα κάνουμε εμείς λοιπόν. Γιατί Πάντα με προβληματίζει αυτό που αναφέρεται σχέση με τους ε, στόχους βιώσιμης ανάπτυξης, ότι ουσιαστικά αναπόκειται στα κράτη-μέλη, αλλά ε, και πάλι τα συζητάμε και με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στον ΟΗΕ. Ξέρετε, ο ΟΗΕ δεν θέλει να λέει στις χώρες τι να κάνουν. Είναι πολύ δύσκολο. Αλλά ακόμα και στην Ευρωπαϊκή Ένωση ε, δεν είναι σαφές ότι θα συλλέξει η Ευρωπαϊκή Ένωση δεδομένα θέλει να παροτρύνει τα κρατημέλη, αλλά δεν λέει θα συγκεντρώσουμε και στοιχεία για να τα συγκρίνουμε, αλλά έτσι θα γνωρίζουμε. Πείτε μας λοιπόν τι θα γίνει στο επίπεδο της παγκόσμιας στρατηγικής, πώς θα στηρίξουμε άλλες χώρες να υλοποιήσουν τον στόχο 16, αλλά να μην ξεχνάμε ότι και η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να τον υλοποιήσει. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ και ζητούμε συγγνώμη και πάλι που η Διευθύντρια Λότε Κνούτσεν δεν μπορούσε να παρευρεθεί. Είμαι εδώ λοιπόν στη θέση της. Θα προσπαθήσω να απαντήσω σε αυτό το ζήτημα και θα αναφερθώ και στην ε, παγκόσμια αυτή στατική για την ε, εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφαλείας που ε, παρουσίασε η Πατή Εκπρόσωπος κ. Μογκερίνη. Θα κάνω και μια μνήα στη σημασία του στόχου και στα ανθρώπινα δικαιώματα και θα σταθώ και στην, στα ευάλωτα σημεία και την αντοχή που είναι κύρια σημεία της παγκόσμιας αυτής ε, στρατηγικής και μερικά ακόμα σημεία για την ευρωπαϊκή στήριξη στο, στη μεταρρύθμιση του τομέα ασφάλειας και στην οικοδόμηση δυναμικού για την ασφάλεια και ανάπτυξη, που είναι λίγο αμφιλεγόμενα ζητήματα αλλά συνδέονται σαφώς με τον SDG 16. Πρώτα απ' όλα συμφωνούμε με τα όσα έχουν αναφερθεί ότι το θεματολόγιο του 2030 αποτελεί πραγματικά μια αλλαγή παραδείγματος εφόσον με την έννοια ότι αποτελεί μια μοναδική ευκαιρία να αλλάξουμε την πολιτική μας και την προσέγγισή μας. Ιδίω για μας την Ευρωπαϊκή Ένωση αφορά και το πώς ε, οι πολιτικές μας, εξωτερική και εσωτερική πολιτική μας θα γίνει ε, πιο συνεκτική ε, και πώς ε, θα συγκεντρώσουμε τις δυνάμεις μας σε επίπεδο κράτων μελών και θεσμικών οργάνων. Η γένεση, όπως αναφέρθηκε προηγουμένως, του στόχου 16, σαφώς και η Ευρωπαϊκή Ένωση διαδραμάτισε πολύ σημαντικό ρόλο για τον προσδιορισμό και την υιοθέτηση του SDG 16 και εν γέννη μπορούμε να πούμε ότι και αυτός ο στόχος, αλλά γενικότερα και όλοι οι στόχοι SDG ε, αντιπροσωπεύουν και τις αξίες ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γι' αυτό ήμασταν πολύ σημαντικός φορέας και στην υλοποίηση, και είμαστε, στην υλοποίηση των στόχων. Αναμένουμε και από τους άλλους εταίρους να είναι ε, και οι ίδιοι στο προσκήνιο αυτής της διαδικασίας και θέλουμε και τα κράτη-μέλη μας να ε, τονίζουν όπως και εμείς ότι ε, μπορούν να κάνουν τη διαφορά αυτή η στόχη. Τώρα αυτή η παγκόσμια στρατηγική που παρουσίασε πριν από μερικούς μήνες ε, η κυρία Μογκερίνη όντως συνδέει, συνδέεται με το θεματολόγιο του 2030 και το ω προτεραιότητα. Πριν από μερικές ημέρες η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 22 Νοεμβρίου υιοθέτησε ένα ε, πακέτο για τη βιώσιμη ανάπτυξη που αποτελεί μια ισχυρή πολιτική δέσμευση και συνεισφορά και την υλοποίηση του θεματολογίου σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επομένω, δεν έχουμε φτάσει ακόμα στο επίπεδο συλλογή και σύγκριση δεδομένων, παρότι υπήρχε στη δέσμη και μία έκθεση τη Eurostat. Όμω, νομίζω τώρα έχουμε ένα σύνολο ε, πολιτικών εντός και εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης για να υλοποιήσουμε το θεματολόγιο 2030. Ο στόχος 16 σαφώς και τη χάνει ευρεία στήριξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση γιατί αναγνωρίζει τη σημασία της ειρήνης, δικαιοσύνης και διακυβέρνηση για τη βιώσιμη ανάπτυξη. Όπως μόλις αναφέρθηκε, ο στόχος αυτός είναι απαραίτητος για να ε, υλοποιηθούν και άλλοι στόχοι. Χρειαζόμαστε λοιπόν αποτελεσματικά θεσμικά όργανα που θα εργάζονται από κοινού ε, με την κοινωνία των πολιτών. Είναι λοιπόν απαραίτητε προποθέσει για την υλοποίηση των στόχων. Δεν γίνεται αλλιώ ε, να ε, πετύχουμε αυτό το στόχο. Απαιτείται μια συμμετοχική προσέγγιση για να έχουμε πραγματικά αποτελέσματα. Και για να γίνει αυτό πρέπει να προωθήσουμε τις πολιτικές χωρίς αποκλισμούς ε, να αυξήσουμε τη συνεργασία μας με την κοινότητα των πολιτών ε, ε, κτλ. Αυτό θα επιτρέψει στην κοινότητα των πολιτών να συμμετάσχει με καλύτερο τρόπο και πιο ενεργό τρόπο στη διακυβέρνηση. Μέσω του SDG 16 η δημοκρατία μπορεί να συμβάλλει για την υλοποίηση πρακτικών αποτελεσμάτων για όλους. Η νέα ευρωπαϊκή κοινή αντίληψη που πρότεινε πριν από μερικέ ημέρε η Επιτροπή ε, τονίζει ότι οι συμπεριληπτικές κοινωνίες και τα υπόλογα θεσμικά όργανα είναι ένα σημείο κλειδί ε, για τη δημοκρατία. Ε, για να αποφύγουμε ε, νέε συγκρούσει και να σταθεροποιήσουμε τι χώρε εταίρου μα, πρέπει να επενδύσουμε στην δημοκρατική διακυβέρνηση που θα οδηγήσει και στην ανάπτυξη, στις νέες θέσεις εργασίας και στη βελτίωση υποδομών όπως είναι η εκπαίδευση και η γενική περίθαλψη. Η Ευρωπαϊκή Ένωση επίσης πάλεψε σκληρά για έναν ε, SDG για τα ανθρώπινα δικαιώματα και ο 16 θα συμβάλλει τα μάλλα ε, στην υιοθέτηση τέτοιων ε, θεματολογίων. Γενικά ακολουθείτε μια σωστή προσέγγιση κατά τη γνώμη μας και διασφαλίστε ότι τα ανθρώπινα δικαιώματα θα εντάσσονται σε οτιδήποτε κάνουμε. Η υποστήριξη της δημοκρατικής κυβέρνηση και ο στόχος 16 όχι μόνο συνάδουν με τις αξίες μας, αλλά ε, ενσωματώνονται και στα συμφέροντά μας. Και η οικουμενική αυτή, η σφαιρική προσέγγιση και στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης επισημαίνει ακριβώς ότι όλα αυτά είναι άρρητα συνδεδεμένα μεταξύ τους. Μάλιστα υπάρχει ένας ε, σαφής σύνδεσμος μεταξύ της ευρωπαϊκής ασφάλειας και των ε, σταθερών ε, ε, γειτονικών χωρών στην ευρύτερη περιφερειά μας. Και έχουμε κατανοήσει ότι όταν είναι δυνατοί οι γείτονές μας, είμαστε και εμείς δυνατοί. Θέλουμε λοιπόν να αντιμετωπίσουμε τις πηγές ε, αστάθειας που οδηγεί χιλιάδες ανθρώπους σε δύσκολους και επικίνδυνους δρόμους. Θεωρούμε ότι ε, η έλλειψη δημοκρατικής διακυβέρνηση είναι μία από τις αιτίε που πρέπει να αντιμετωπίσουμε και το Ευρωπαϊκό Εξωτερικό Σχέδιο Επενδύσεων, το οποίο τώρα εξετάζει και το Συμβούλιο και σύντομα και το Κοινοβούλιο, έχει υποβληθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση σε αυτό το πλαίσιο ανάπτυξη τη νέα κοινή αντίληψη για την ανάπτυξη και για την βιώσιμη ανάπτυξη ευρύτερα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θέλει να ακολουθήσει μια τέτοια σφαιρική προσέγγιση για την αποτροπή αυτών των κρίσεων. Θέλουμε λοιπόν μεγαλύτερη συνοχή, ιδίω στου τομεί τη μετανάστευση, του εμπορίου και των επενδύσεων, αναπτυξιακή συνεργασία και καταπολέμηση τη τρομοκρατία. Η Ευρωπαϊκή Ένωση υιοθέτησε περάσματα του Συμβουλίου για την ε, προσέγγιση αυτή για την αναπτυξιακή συνεργασία το 2014. Τώρα, σε ό,τι αφορά τις ε, αδυναμίες, τα τροτά σημεία και την ανθεκτικότητα. Υπάρχουν μεγάλες ε, ανισότητες στον κόσμο και αυτά ε, οδηγούν σε αστάθεια και συγκρούσεις. Πολλές από αυτές τις συγκρούσεις ε, λαμβάνουν χώρα σε τέτοιες αδύναμες, σε βάλλοντες χώρες και η ανασφάλεια αυτή οδηγεί σε χαμηλότερες επενδύσεις και περαιτέρω φτωχοποίηση. Με τη στρατηγική μας λοιπόν δίνουμε μεγάλη έμφαση στην ε, ανθεκτικότητα, η αντοχή, δηλαδή τη δυνατότητα ε, ταχείας ε, ανάκαμψης και αποτροπής μελλοντικών κρίσεων. Συνδέεται με τις καλές θέσεις εργασίας και την ανάπτυξη, με ίσες ευκαιρίες για όλους, πέραν του φύλου, των θρησκευτικών πεπιθήσεων ή της εθνικότητας. Όμως, ε, συνδέεται και με το κράτο δικαίου, τη δικαιοσύνη και τη διαβούλευση. Συνδέεται λοιπόν άμεσα με τον SDG ε, 16. Θέλουμε να εξετάσουμε την αντοχή κρατών και κοινωνιών ε, για να αντιμετωπίσουν εσωτερικές εντάσεις και να ανακάμψουν μετά από κάποιους κρατασμούς. Έτσι θα έχουμε περισσότερη ειρήνη και ευημερία στον κόσμο και η συσχέτιση μεταξύ δημοκρατίας, ασφάλειας και ευημερίας θα οδηγεί σε καλύτερα αποτελέσματα και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στις εξωτερικές, στις διεθνείς τη σχέσεις. Θέλουμε επίσης να ενισχύσουμε την ευρωπαϊκή διαχείριση ε, κρίσεων και συγκρούσεων, εμβαθύνοντα το έργο μας ε, μέσω μιας ολοκληρωμένη προσέγγισης που θα λαμβάνει υπόψη ε, όλες τις διαστάσεις των συγκρούσεων αυτών. Έτσι θα ενισχύσουμε την συνοχή των ευρωπαϊκών ε, ε, απαντήσεων σε τέτοιες περιπτώσεις ε, κρίσεων και συγκρούσεων με στόχο την εξέβρεση λύσεων. Τώρα, σε ό,τι αφορά την μεταρρύθμιση στον τομέα της ασφάλειας, θεωρούμε ότι το να στηρίξουμε φορείς του τομέα της ασφάλειας είναι απαραίτητο στοιχείο για να διασφαλίσουμε ότι υπάρχουν οι απαραίτητες προϋποθέσεις για την ασφάλεια και τη σταθερότητα. Έτσι, το Συμβούλιο στις 14 Νοεμβρίου υιοθέτησε ένα νέο στρατηγικό ε, πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για αυτόν τον σκοπό. Αυτό το νέο πλαίσιο πολιτικής, το οποίο συμμερίζονται όλοι οι φορείς, ε, θα μας δώσει δυνατότητα να παράσχουμε ολοκληρωμένη στήριξη σε χώρε εταίρου στην προσπάθειά τους να βελτιώσουν τη διακυβέρνηση του τομέα ασφάλειάς τους και στις ικανότητές τους ε, να ανταποκρίνονται στις ε, ε, ανάγκες ασφάλειας του πληθυσμού τους. Όλοι γνωρίζουμε ότι μία νομιμοποιημένη ε, υπόλογη υποδομή ω προ την ασφάλεια είναι ένα απαραίτητο στοιχείο γενικότερα και θα βοηθήσει και την Ευρωπαϊκή Ένωση να διασφαλίσει την ασφάλειά τη και εντό και εκτό των συνόρων τη. Αυτό το νέο πλαίσιο πολιτική θα συμβάλλει και στου ε, κεντρικού στόχου της Ευρωπαϊκής Ένωσης τη ε, προαγωγή ε, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, τη δημοκρατία και της βιώσιμης ανάπτυξη, αλλά και του στόχου της σταθερότητας και της ειρήνης. Με αυτό το νέο πλαίσιο πολιτική, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η Υπηρεσία Εξωτερική Δράσης επίσης σημειώνουν πρόοδο σε ό,τι αφορά την οικοδόμηση δυναμικού, σε ό,τι αφορά την ασφάλεια. Αυτό που ε, μια πρωτοβουλία γνωστή ως CBSD. Θέλουμε να τροποποιήσουμε το μέσο που συμβάλλει στην ασφάλεια και ειρήνη ε, και να συμπερι... σταθερότητα και ασφάλεια και για να συμπεριλάβουμε και τον ε, τομέα της ασφάλειας, ιδίως σε συγκεκριμένε ε, περιπτώσεις. Και αυτό θα συζητηθεί ε, σύντομα και με το Κοινοβούλιο. Είναι σημαντική αυτή η πρωτοβουλία για να υλοποιήσουμε τον στόχο 16 και για να καλύψουμε ένα κενό σε ό,τι αφορά την αποδοτικότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης να στηρίξει τον τομέα ασφαλείας χωρών εταίρων. Οι φορείς ε, ε, που ασχολούνται με το ζήτημα της ασφάλειας, όπως οι ενόπλες δυνάμεις, ε, σε κάποιες ευάλωτες αποσταθεροποιημένες χώρες μπορούν να συμβάλλουν στην ασφάλεια και να διαμορφώσουν τις συνθήκες για την βιωσιμότητα. Η πρότασή μας λοιπόν προβλέπει τέτοια στήριξη να μπορεί να χορηγηθεί σε έκτακτες περιπτώσεις, σε συμφωνία με την χώρα εταίρο και ε, σαν λύση τελευταίας ανάγκης σε περίπτωση ε, απειλών για την δημοκρατική λειτουργία των θεσμών και της ασφάλειας. Δεν υπάρχουν άλλες καλύτερες επιλογές για να φέρουμε την ε, ασφάλεια και σταθερότητα στον κόσμο. Και αυτή η στήριξη θα είναι και μια ευκαιρία να βελτιώσουμε τη διακυβέρνηση ε, και λογοδοσία αυτών των φορέων. Επιβεβαιώνω λοιπόν ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση αποδίδει ιδιαίτερη σημασία στην υλοποίηση του SDG 16. Είναι σημαντικό τα θεσμικά όργανα και τα κρατημέλη να συμμετέχουν όλο και περισσότερο από κοινού ε, και στο όραμα τους και ε, πρακτικά για να ενισχύσουν τη φωνή της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον κόσμο. Σας ευχαριστώ πολύ. Um, um, Σας ευχαριστούμε ε, πολύ. ακούσαμε τις σχέσεις αυτές με την και θα ακούσουμε τώρα από τον Ζαν Λουί Βιλ, τον οποίο έχουμε προσκαλέσει και στο παρελθόν επανειλημμένα και θα θέλαμε να ακούσουμε από τον ε, συνάδελφο Βιλ ε, ε, το τι ακριβώ θα πρέπει να αναμένουμε από αυτήν την αντίληψη. Είχαμε δηλαδή την μέχρι τώρα την αντίληψη, αλλά τι ακριβώς να, να αναμένουμε από τον στόχο 16, το στόχο βιώσιμη ανάπτυξη 16 στο πλαίσιο της νέα κοινή αντίληψη. Ποια θα είναι τα νέα στοιχεία, τι θα αλλάξει. Αυτό είναι το ερώτημα που θέτω. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ελπίζω πως πράγματι θα υπάρξει αλλαγή. Αυτή είναι η σύντομη απάντηση που μπορώ να σας δώσω. Καταρχήν ε, να σας ευχαριστήσω σε κάθε περίπτωση για την πρόσκλησή σας να συμμετάσχω σε αυτό το πάνελ και θα προσπαθήσω να απαντήσω στα ερωτήματα που μας θέσατε χωρίς να επαναλάβω τα όσα είπαν ε, πριν από μένα οι συνάδελφοι. Γιατί ήδη βέβαια αναφέρθηκαν στα επιχείρηματα υπέρ της, του οικονομικού χαρακτήρα και της διασύνδεσης του ε, στόχου SDG 16 με τους υπόλοιπους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης. 1, 4, 5, δηλαδή ε, παιδεία, φτώχεια ε, και ισότητα φύλων είναι και αυτοί οι στόχοι οι οποίοι σχετίζονται με, το έργο μας ε, σε αυτό το πλαίσιο. Τώρα, σε ό,τι αφορά ε, το, την ατζέντα του 2030. Ο στόχος βιώσιμης ανάπτυξης 16 είναι ιδιαίτερα σημαντικός. αλλά δεν νομίζω, αν και δεν υποτίθεται πως πρέπει να πω κάτι τέτοιο, ότι θα αποτελέσει τον παράγοντα που θα επιφέρει την αλλαγή. Ναι, έχουμε 15 χρόνια μπροστά μας για να επιτύχουμε κάποιες αλλαγές, αλλά είμαστε ταυτόχρονα και ρεαλιστές. Ε, και νομίζω πως και η Σάρα το ανέφερε, με σαφήνει αυτό. Δηλαδή, ας μην υποτιμούμε ε, τις διαστάσεις ε, των προκλήσεων ε, που αντιμετωπίζουμε. Και ο Φελιμπέρτο αναφέρθηκε σε αυτό ότι δηλαδή την περασμένη εβδομάδα η Επιτροπή ε, υιοθέτησε ένα νέο πακέτο ε, για αυτόν τον πυλώνα με την, το μέλλον για την Συμφωνία Κουτουνού όπου υπάρχει ακριβώς και αυτή η γενική εφαρμογή των στόχων της βιώσιμης ανάπτυξης. Και βέβαια ε, έχουμε και τη νέα κοινή αντίληψη η οποία ε, προτείνεται σε ανακοίνωση της Επιτροπής σε ό,τι αφορά ε, την ανάπτυξη και έτσι έχουμε αυτά τα βασικά στοιχεία με βάση τα οποία θα δομήσουμε την προσέγγιση μας απέναντι στην επίτευξη των στόχων SDG. Νομίζω πως μέσω πολιτικού διαλόγου και αναπτυξιακής συνεργασίας θα επιτύχουμε τη συνεργασία μεταξύ όλων των εταίρων, δηλαδή μεταξύ μόνο των κρατώμενων αλλά και των υπολείπων χωρών προκειμένου να επιτύχουμε ακριβώς αυτούς τους ε, οικονομικούς ε, στόχους, ε, δηλαδή η εξάλληψη τη φτώχεια, η προώθηση της δημοκρατική διακυβέρνησης, η διατήρηση της ειρήνης. Τώρα, από εκεί και μετά σε ό,τι αφορά την αναπτυξιακή συνεργασία και τη σχετική χρηματοδότηση, γιατί βέβαια συχνά αυτό είναι το ζήτημα για το οποίο δίνεται προσοχή σε εμά. Να πω ότι δεν είναι πάντοτε το πιο σημαντικό ζήτημα τη χρηματοδότηση. Το σημαντικό είναι να γίνουν οι σωστέ επιλογέ. Και ποιε είναι αυτέ οι επιλογέ που θα κληθούμε να κάνουμε. Ε, θα είδατε στη νέα κοινή αντίληψη για την ανάπτυξη, γιατί φαντάζομαι ότι όλοι σα θα τη διαβάσατε και θα ξέρετε απ' έξω. Θα είδατε λοιπόν σε, σε αυτό το νέο consensus ότι εστιάζουμε σε αυτά τα 5P, σε αυτές τις 5 διαστάσεις, 5P ε, τα λέμε στα αγγλικά για να τα θυμόμαστε εύκολα, δηλαδή people, άνθρωποι, planet, πλανήτης, prosperity, ευημερία, peace, ειρήνη και partnership, εταιρική σχέση. Έτσι θα προσπαθήσουμε λοιπόν να, να χωρίσουμε αν θέλετε σε επιμέρους στοιχεία το σύνολο αυτού του στόχου. Και πώς λοιπόν τώρα θα συνδέσουμε αυτή την κοινή ε, αντίληψη για την ανάπτυξη με τον στόχο 16. Όπως είπαμε κυρία Πρόεδρε, δεν ξεκινάμε από το 0 και αυτό ε, το ανέφερε και η Σάρα κατά την παρουσίασή της όταν είπε δηλαδή ότι ήδη έχουμε πολύ αρκετή εμπειρία ε, από άλλους αναπτυξιακού στόχου τη χιλιατίας η οποία δεν ήταν αμυγός στόχη σε ό,τι αφορά την διακυβέρνηση. Αλλά ε, ε, σίγουρα ε, σε ό,τι αφορά για παράδειγμα τους στόχους για την αλλαγή ένας από τους δύο πυλώνες ήταν πάντοτε η διακυβέρνηση και έχουμε λοιπόν εφαρμόσει προγράμματα σε ό,τι αφορά την προώθηση της χρηστή διακυβέρνησης σε ένα μεγάλο αριθμό κρατών τόσο κρατών, δηλαδή τόσο σε κράτη όπου υπάρχει μακρά παράδοση σταθερότητας όσο και σε κράτη τα οποία πρόσφατα έχουν βγει από περίοδο κρίσης ε, όπως εσείς τα γνωρίζετε και σας το συγγνώμη αν επαναλαμβάνω πράγματα που ήδη γνωρίζετε, ε, σε 70 ε, χώρες ήδη η διακυβέρνηση αποτελεί ένα από τα focal sectors, δηλαδή από τους τομείς στους οποίους ε, εστιάζουν. Από δηλαδή από 110-120 χώρες, πάνω από το ίμιση, 70 δηλαδή χώρες, έχουν στο πλαίσιο της διμερούς συνεργασίας ως ένα από τα θεματικά πεδία τη διακυβέρνηση. Και χρησιμοποιούμε λοιπόν όλους τους ε, δυνατούς ε, διάβλους ε, που έχουμε στη διάθεσή μας για να επιτύχουμε αυτή την αλλαγή, δηλαδή και σε επίπεδο των δημοσιοκυβερνήσεων όπως και στο επίπεδο ιδιωτικών επιχειρήσεων, οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών, περιφερειακό επίπεδο και ούτω καθεξής, δεν χρειάζεται να τα επαναλάβω. Και εδώ έχουμε ένα μείγμα όλων αυτών των προσεγγίσεων. Δεν υπάρχει δηλαδή μια ενιαία προσέγγιση την οποία εφαρμόζουμε από την πλευρά τη Ευρωπαϊκή Ένωση απέναντι σε όλου. Κάθε χώρα είναι διαφορετική, ε, κάθε πλαίσιο είναι διαφορετικό ε, και κάθε φορά οι παράγοντε αλλαγή μια χώρα είναι διαφορετικοί. Οπότε θα πρέπει να παραμείνουμε ευέλικτοι, θα πρέπει να και θα πρέπει πάντοτε να λαμβάνουμε υπόψη μας τις τοπικές ιδιαιτερότητες της κάθε χώρας ε, δηλαδή. Ε, και αυτό όταν, ε, σε ό,τι αφορά την επιλογή των εργαλείων μας, σε ό,τι αφορά τη χρηματοδότηση, σε ό,τι αφορά την, την επιλογή των καταπιστευματικών ταμείων και ούτω καθεξής. Και εδώ έχω δύο παραδείγματα χωρών. Την Πενίνη, η οποία σίγουρα δεν είναι χώρα η οποία διέρχεται κρίση, αλλά πρόκειται για μια χώρα στην οποία έχουμε εμπλάκει ε, για να προωθήσουμε την ε, δημοκρατική διακυβέρνηση σε ένα σταθερό πολιτικό περιβάλλον. Μέσα σε μερικές εβδομάδες θα ξεκινήσει η Επιτροπή ε, μια μαζική χρηματοδοτική ενίσχυση της τάξης των 83 εκατομμυρίων ευρώ στον τομέα ακριβώ τη διακυβέρνηση και δεν είναι αμεληταίο αυτό το ποσό και θέλουμε να αποτελέσει ένα μοχλό για να επιτύχουμε διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις και να μειώσουμε τα εμπόδια απέναντι στην ατιμορρησία, δηλαδή αυτό στο επίπεδο της ε, δεδομένης της ε, μετά να ενισχύσουμε τις ε, κρατικές αρχές, να αυξήσουμε και τη διαφάνεια του εθνικού φορολογικού συστήματος. Άρα λοιπόν αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε είναι να ανταποκριθούμε σε μία σειρά από διαφορετικά ζητήματα σε κάθε χώρα. Είτε αυτά αφορούν για παράδειγμα το φορολογικό σύστημα, είτε αφορούν ε, το, τη δικαιοσύνη, είτε αφορούν το ευρύτερο θεσμικό πλαίσιο. Δηλαδή δεν έχουν να κάνουν μόνο με ένα τομέα, για παράδειγμα μόνο το Υπουργείο Δικαιοσύνη μια χώρα ή κάτι άλλο. Κάτι το οποίο είναι αξιοσημείωτο και θα ήθελα να το τονίσω εδώ, είναι ότι η εν λόγω επιχείρηση αυτή τη στιγμή ξεκίνησε ε, ε, ε, με βάση μια ανάλυση της κρατικής ακαιρεότητας ε, της Μενλίν που έλαβε χώρα από την Transparency International. Δηλαδή διαπιστώθηκε ακριβώς, ε, έγινε με διαπίστωση ό,τι αφορά την κατάσταση σχέση με την ε, διάφθορα σε αυτή τη χώρα και μετά έγινε και με τη συνεργασία των αρχών της Μενλίν. Οπότε έχουμε ένα από τα πιο σημαντικά στοιχεία τα οποία είναι απαραίτητα για να στεφτεί με επιτυχία μια τέτοια προσπάθεια, δηλαδή την εμπλοκή ή την, την, την θετική στάση των ε, κρατικών αρχών. Ε, και προφανώς ε, προσπαθούμε σε αυτό το πλαίσιο να ενισχύσουμε και το πολιτικό διάλογο σε ό,τι αφορά τη, τη διαφθόρα. Τώρα, ένα εντελώ διαφορετικό πλαίσιο. Πριν από δύο εβδομάδε έλαβε χώρα εδώ στι Βρυξέλλε μια μεγάλη διάσκεψη σε ό,τι αφορά την κεντρική Αφρικανική Δημοκρατία. Και εδώ έχουμε ένα εντελώ αντίθετο παράδειγμα προ αυτό τη Μπενίν. Δηλαδή έχουμε ένα σταθέ κράτο το οποίο μόλι τώρα εξέρχεται από μια ένοπλη σύραξη, έχουμε κοινότητες οι οποίες έχουν διαραγεί, έχουν, βρίσκονται σε σύραξη μία ε, με την άλλη από το 2015 ε, και αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε είναι καθ' όλη τη διάρκεια της κρίσης να παρέχουμε υποστήριξη ε, μέσω για παράδειγμα αποστολών ανθρωπιστικής βοήθειας και μέσω όλων των εργαλείων που έχουμε στη διάθεσή μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση ώστε να σταματήσει καταρχήν η ένοπλη σύραξη και από εκεί και μετά να ξεκινήσει πάλι η ε, διαδικασία σταθεροποίησης ε, και διαδικασία του να καταστεί και πάλι αποτελεσματικό και έβρισμα λειτουργών το κράτο. Ε, δημιουργήσαμε ένα καταπληκτικό ταμείο με την ονομασία Μπεκού που περιλαμβάνει ακριβώς τα ζητήματα αποκατάστασης και ανοικοδόμησης, ξεκινώντας δηλαδή ακριβώς από αυτήν την διαδικασία μετάβαση από την κρίση στην σταθερή κατάσταση και εδώ έχουμε να κάνουμε δηλαδή και με την κοινωνία των πολιτών, την ασφάλεια της, ε, των, ε, της διατροφικής αλυσίδας και ε, την, επίσης την υποστήριξη του, της δίκαιας της νομίμου εκλογικής διαδικασίας και της διαφάνειας αυτή τη διαδικασία. Όμως αυτό προσπαθούμε να κάνουμε μετά ακριβώς από την οξία περίοδο της διαχείρισης της κρίσης είναι να προβούμε σε μια αξιολόγηση, αποκοινούμε και τη Δυτική Αφρικανική Δημοκρατία προκειμένου να ε, καταρτιστεί ένα ε, ε, σχέδιο δράση για την ανοικοδόμηση και την ειρηνευτική διαδικασία, το οποίο παρουσιάστηκε σε αυτή τη διάσκεψη πριν από δύο εβδομάδε εδώ στι Βρυξέλλε. Αυτό καταδεικνύει την ανάγκη να υπάρξει περαιτέρω συνεργασία, αν θέλετε, σε ό,τι αφορά την περαιτέρω αναπτυξιακή υποστήριξη και την ανθρωπιστική βοήθεια. Τι προσπαθώ να σας πω με αυτά τα δύο παραδείγματα που σας ανάφερα. Θα πρέπει να έχουμε κατά νου ότι η φτώχεια θα συνεχίσει να συγκεντρώνεται ιδιαίτερα στις χώρες εκείνες οι οποίες πλήττονται από πολέμους και από πολιτική αστάθεια. Και αυτό το διαπιστώνουμε και ε, με βάση τις ε, προβλέψεις για τις χώρες οι οποίες βρίσκονται σε μια τέτοια ασταθή κατάθεση. Το 43% λοιπόν, ε, του πληθυσμού που πλήττεται σε αυτές τις χώρες από αυτή την αστάθεια θα έχει αυξηθεί στο 62%. και ε, παρότι δεν μπορώ να σας αναφέρω τώρα ακριβώς ε, ε, την πηγή, σίγουρα καταδεικνύει μια τάση που βλέπουμε. Αν λοιπόν θέλουμε πραγματικά να ξαλείψουμε, τουλάχιστον να μειώσουμε την τότε σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να συνεχίσουμε να βελτιώνουμε τις μεθόδους εργασίας μας σε ό,τι αφορά την ενίσχυση της πολιτικής σταθερότητας και αυτή είναι και η μόνη άγουσα την οποία μπορούμε να ακολουθήσουμε. Δηλαδή βιώσιμη ανάπτυξη. Σε διαφορετική περίπτωση δεν δεν θα κάνουμε τίποτα άλλο παρά να προωθήσουμε ένα σύστημα το οποίο τελικά δεν θα είναι βιώσιμο μακροπρόθεσμα. Ε, θα χρησιμοποιήσουμε την ίδια συνταγή, αν μπορώ να την πω έτσι, εντό εισαγωγικών, γιατί δεν μου αρέσει πολύ αυτή η έκφραση. Προσπαθούμε σε κάθε περίπτωση να ακολουθήσουμε την ίδια προσέγγιση που ακολουθήσαμε και στην κεντρική Αφρικανική Δημοκρατία στο κέρα της Αφρικής, ε, για παράδειγμα στις χώρες της Σαχέλ ή στη Νότια Ασία. Μπορούμε να έχουμε να κάνουμε περιοχές όπου μπορούμε να ακολουθήσουμε αυτή την προσέγγιση. Επιτρέψτε μου ε, πάντως κλείνοντας να αναφερθώ σε τρία ζητήματα. Η ε, ευαισθησία σε σχέση με τις συγκρούσεις, η αστάθεια δηλαδή με βάση τις συγκρούσεις είναι πάρα πολύ σημαντική και σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να τη λάβουμε υπόψη μας. Ε, δηλαδή θα πρέπει ε, να το κατανοήσουν αυτό όλοι στο δικό μας επίπεδο του προσωπικού μας ε, και να το προσεγγίσουν όλοι γιατί σε διαφορετική περίπτωση η δική μας παρέμβαση δεν θα έχει τον αντίκτυπο που θα μπορούσε να έχει και ενδεχομένως να αποδειχθεί και επιζήμια αντί ε, να ενοφέλουμε. Δεύτερο, σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να δράσουμε από κοινού. Και το γεγονό, για παράδειγμα, το ότι έχουμε έναν εκπρόσωπο ε, των Ηνωμένων Εθνών σε αυτό το πάνελ καταδεικνύει το, την ανάγκη αυτή τη συνεργασία. Ε, δεν θα πρέπει να επιλέξουμε δηλαδή τον έναν ή τον άλλον. Ε, δεν μπορούμε να δράσουμε απομονωμένα ο καθένας πρεσβεύοντας δηλαδή με βάση τη δική του σημαία εκείνα τα οποία νομίζει πως είναι σωστά χωρίς να λαμβάνει υπόψη ε, τους άλλους και χωρίς να τους συμπεριλαμβάνει σε αυτή την προσπάθεια. Και τρίτο σημείο που θα ήθελα να τονίσω είναι ότι θα πρέπει να επενδύσουμε σε μεγάλο βαθμό στην ε, ε, πρόληψη των ε, συγκρούσεων και στην ευτική διαδικασία και στην διατήρηση του κράτους σε δικαίου. Και ο Λιμπέρτο αναφέρθηκε ακριβώς στην προσέγγιση που ακολουθείται και από την πλευρά των ΗΠΑ και αυτό θα αποτελέσει και για μας ένα βασικό στοιχείο των εργασιών μας. Κλείνοντας ή συνοψίζοντας, θα πρέπει λοιπόν να ε, ε, ενισχύσουμε την ε, ασφάλεια, την ανθεκτικότητα των κρατικών μηχανισμών, τις οικονομικές ευκαιρίες οι οποίες βέβαια είναι απαραίτητες για να διατηρηθούν αυτά τα επιτεύγματα. Άρα λοιπόν όλα αυτά είναι απαραίτητα, ναι, αλλά ο στόχος SDG 16 θα αποτελέσει πραγματικά το θεμέλιο, αν θέλετε, για το οποίο θα κρίνει και την επιτυχία μας στους υπόλοιπους στόχους. Μαρία, μόνο οι επίγουσες ερωτήσεις παρακαλώ, γιατί δεν έχουμε χρόνο. Μία παρατήρηση μόνο θέλω να κάνω. δεν μπορώ ακριβώς να φανταστώ πώς θα εφαρμοστεί αυτό το στόχο στην ε, πράξη. Δεν ξέρω αν ακούτε καλά. Άλλος δεν μπορώ λοιπόν να φανταστώ πώς θα εφαρμοστεί αυτός ο στόχος ε, στην πράξη, γιατί βέβαια όλοι αυτοί οι στόχοι συνδέονται και εξαρτώνται ο ένας από τον άλλον, οπότε θα είναι περίπλοκη αυτή η διαδικασία και είναι σημαντικό να ε, αναπτύξουμε και τους κατάλληλους δείκτες για να μετρήσουμε την επίδευξη αυτών των στόχων. Ε, και άκουσα τη συνάδελφο που είπε ότι, ότι καλούνται τα κράτη-μέλη να εφαρμόσουν αυτούς τους στόχους. Ε, ναι, μεν θα πρέπει να αναλάβουν τις ευθύνες τους τα κράτη μελά και τα κράτη γενικά που συμμετέχουν, αλλά όλοι οι αρμόδιοι φορείς θα πρέπει να αναλάβουν τις δικές τους ευθύνες για την επίτευξη αυτών των στόχων και αναφέρομαι σε όλα τα επίπεδα, μέχρι και στο επίπεδο των Δήμων και Κοινοτήτων. αναφερθήκα σε αυτά τα πέντε ε, άνθρωποι, πλανήτης, ε, ευημερία, ειρήνη εταιρική ε, σχέση. Προφανώς αυτά τα ζητήματα θα πρέπει να, παίξουν, να έχουν την κατάλληλη πολιτική βαρύτητα σε όλα τα επίπεδα διακυβέρνηση και στα, ε, στις ε, χώρες, δηλαδή ξεκινώντας από τους Δήμους και τις κοινότητες και φτάνοντας μέχρι στους διεθνείς οργανισμούς, στα Ενωμένα Έθνη, για να υπάρξει πραγματικά επιτυχία. Αφού πρόκειται για τόσο γενικούς στόχους. Οπότε η δική μου αίσθηση είναι ότι δεν είμαστε ακόμα έτοιμοι για να ελέγξουμε όλους τους, ε, όλα τα πεδία πολιτικής και επίσης δεν έχω ακούσει μια ιδέα ως προς το πώς θα προσεγγίζουμε συστηματικά την επίτευξη αυτών των στόχων. Θα πρέπει να είναι πολύ συστηματική η προσέγγιση μας σε ό,τι αφορά όλους τους επιμέρους κλάδους. Ε, για παράδειγμα στη Γεωργία στον κλάδο τη γεωργία. Ε, εγώ μπορώ να σκεφτώ μόνο το τι μπορεί να συμβεί στην, στην Γερμανία, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά για παράδειγμα, αν πούμε ότι εμεί θα βασιστούμε στι εξαγωγέ σε κρέατο ποιον αντίκτυπο θα έχει ε, κάτι τέτοιο. Ε, όταν για παράδειγμα εμείς θέλουμε να αποκτήσουμε πρόσβαση σε μια γεωργική αγορά άλλη χώρα και για να γίνει κάτι τέτοιο θα πρέπει να αλλάξει η νομοθεσία σε εκείνη τη χώρα. Τι θα σημάνει αυτό για αυτή τη χώρα σε επίπεδο αναπτυξιακό. Αυτά θα πρέπει να σκεφτούμε. Ευχαριστώ. Πρόεδρε, θα ήθελα καταρχήν να, να ευχαριστήσω τους ομιλητές για αυτές τις παρουσιάσεις. Κράτησα και πολλές ε, σημειώσεις. Ακούσαμε και ε, σήμερα το πρωί την παρουσίαση των ανακοινώσεων της Επιτροπής. Πρόκειται για κάτι ε, πολύ σημαντικό και ε, εγώ και ο, ο συνάδελφος Νόιζερ ε, προετοιμάζουμε αυτή την περίοδο μια σχετική γνωμοδότηση Και σε αυτή τη γνωμοδότηση πράγματι ε, διαπιστώνουμε και εμείς ε, πως ε, η κοινή αντίληψη παίζει πολύ σημαντικό ρόλο σε διάφορους ε, τομείς όπως για παράδειγμα του, του περιβάλλοντος των τροφίμων και άλλων. Αναφέρθηκε και το ζήτημα βέβαια της ε, ασφάλειας σε διάφορα επίπεδα και των τοπικών αρχών. Αναφερθήκαμε και αναφερόμαστε και στην έκθεση στις συνδικαλιστικές οργανώσεις, στις ενώσεις των οργοδοτών αλλά σε κάθε περίπτωση συνεργασία και επικοινωνία είναι πολύ σημαντικά στοιχεία. Το ερώτημα όμως που τίθεται είναι ε, ποιο θεωρείται πως θα είναι ο ρόλος που θα παίξουν τα εθνικά κοινοβούλια. Δηλαδή όταν λέμε στόχος SDG 16 εννοούμε ότι θέλουμε να υπάρχουν ισχυρά κρατικά θεσμικά όργανα. Και μπορεί να είναι γενικός αυτός ο στόχος, στη διατύπωσή του, αλλά σίγουρα θα χρειαστεί από εκεί και μετά να συγκεκριμενοποιηθεί και χρειαζόμαστε και το άλλο χρόνο για να ξεκινήσει η συνεργασία μεταξύ των αρμόδιων φορέων, προκειμένου πράγματι να επιτύχουμε τελικά την ύπαρξη τέτοιων ισχυρών θεσμικών οργάνων. Και αναφέρθηκε ήδη, για παράδειγμα, ε, το ζήτημα του κράτου δικαίου και τη ενίσχυση του τομέα τη δικαιοσύνη. Επίση, θα ήθελα να αναφερθώ στο ε, σχέδιο εξωτερικών επενδύσεων τη Ευρωπαϊκή Ένωση εδώ έχουμε μια εταιρική σχέση την οποία συζητάμε αυτή την περίοδο και θα ήθελα να σας ρωτήσω πώς ακριβώς θα διαμορφωθεί ε, θα διαμορφωθεί αυτό το σχέδιο εξωτερικών επενδύσεων σε σχέση με τις χώρες της Αφρικής. Πώς θα μπορούσαμε δηλαδή να αξιοποιήσουμε αυτό το σχέδιο για να επωφεληθούν και οι μικρότερες επιχειρήσεις. Γιατί βέβαια και με τέτοιου είδους εργαλεία προς μικρές επιχειρήσεις ενισχύουμε και τις ε, τοπικές αγορές. Εργασίας. Ας ξεκινήσουμε αντίστροφα. Αλλά θα πρέπει να απαντήσετε γρήγορα. Δεν έχουμε πολύ χρόνο. Ζωνα Λουί, να απαντήσει πρώτος. Και οι υπόλοιποι ας προσθέσουν κάτι μετά από σένα. Ο Ζωνα Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Σύντομα. Για να αφήσω περιθώριο στου συναδέλφου να μιλήσουν κι αυτοί. Στην πρώτη ομιλήτρια ε, σίγουρα είναι πολιτική για την ανάπτυξη και κάπου εντάξει συνθήκη, δεν θυμάμαι πού τώρα. Ε, δεν θυμάμαι το άρθρο το συγκεκριμένο, αλλά έχετε πολύ το δίκιο. Εάν δεν είμαστε συνεπείς σε σχέση με αυτά που λέμε και αυτά που κάνουμε, ε, δημιουργούμε, δημιουργούμε πρόβλημα. Θα απαντήσω πολύ σύντομα. Το θέμα ξέρετε ότι όμως είναι τεράστιο αυτό που έκανε η Κομισιόν την προηγούμενη εβδομάδα το έκανε για να υπάρχει συνέπεια. Δηλαδή, ξέρετε ότι ό,τι κάνουμε στην ε, γεωργία έχει επιπτώσει αλλού. Αυτό δεν είναι ξεκάθαρο σε όλου. Το θέμα δεν το λέμε μόνο. Το θέμα είναι να δημιουργήσουμε και ένα σχέδιο και να προχωρήσουμε προ αυτήν την κατεύθυνση. Γιατί αλλιώ ε, θα συνεχίσουμε με τον ίδιο τρόπο. Για κάποιου τομεί αυτό είναι πιο σαφέ. Ε, κλιματική αλλαγή, περιβάλλον, είναι ξεκάθαρο αυτό. Ε, το έχει καταλάβει το κοινό γενικά, η κοινή γνώμη. Ότι ό,τι κάνουμε εδώ στην Ευρώπη μπορεί να έχει επίπτωση στο τι συμβαίνει στον πλανήτη. Μερικές φορές για το εμπόριο ισχύει, για τη γεωργία. Ε, απλώς αναφέρω δειγματοληπτικά κάποια. Μην ξεκινήσω τώρα μία διαφωνία έτσι. Για το επενδυτικό σχέδιο, η εταιρική σχέση με την Αφρική και πώς ε, μπορούμε να βελτιώσουμε τις μικρομεσαίες τις μικρές συγγνώμη, επιχειρήσεις. Δεν ξέρω 100% πώς να το κάνουμε. Δεν πρέπει να εστιάζουμε μόνο στις μεγάλες εταιρείες, αλλά και στις μικρές. Γιατί η, στην Αφρική, όπως και αλλού, η δημιουργία θέσεων απασχόλησης ε, γίνεται και εξασφαλίζεται και χάρη στις μικρές επιχειρήσεις. Υπάρχουν κάποια σχήματα για την ενέργεια που προσπαθούμε να προωθήσουμε έργα μικρής κλίμακας ε, υποστήριξη μικρής κλίμακας, ε, να υποστηρίξουμε δηλαδή τις μικρές επιχειρήσεις στον τομέα της ενέργειας και κυρίως των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Αλλά τώρα δεν σας απαντάω σφαιρικά, σας απαντάω μόνο για τον τομέα, για την ενέργεια. Θα μπορούσα να σας δώσω συμπληρωματικά και άλλες λεπτομέρειες ε, αργότερα. Ο επόμενος ομιλητής, πολύ σύντομα. Ευχαριστώ Πρόεδρε, να εστιάσω κυρίως σε αυτά που ακούσαμε για το ρόλο των κοινοβουλίων. Υποστηρίζουμε τη δουλειά για την ε, υποστήριξη της δημοκρατίας. Το Κοινοβούλιο και συνεργάζεται με τα δικά μας θεσμικά όργανα. Να χρησιμοποιήσουμε όλη τη γνώση, όλες τις συστάσεις που απορρέουν από τις αποστολές ε, εκλογικής, ε, παρατήρηση των εκλογικών αναμετρήσεων εγώ είχα πάει στην ε, Τανζανία, ήμουνα στην Τανζανία πριν πρόσφατα και υποστηρίζαμε το, το, κοινοβούλιο της Τανζανίας ή της Ζανζιβάρης. Ε, εκεί ήρθε η δική σας αποστολή. Ε, τέτοιες ε, προσπάθειες θα πρέπει να τις επεκτείνουμε. Είναι πολύ σημαντικό να υπάρχει αυτή η συμμετοχή ε, που εντάσσεται στο στόχο SDG 16. Για το επενδυτικό σχέδιο, το εξωτερική του διάσταση. Με το επενδυτικό σχέδιο θέλουμε να αυξήσουμε το επίπεδο των χρηματοδοτικών κινήτρων που δίνονται σε επιχειρήσεις ή στα χρηματοδοτικά ιδρύματα για να επενδύσουν σε χώρες που κανονικά δεν προσελκύουν τέτοιους επενδυτές. Για να καλύψουμε και τις ε, προβληματικές χώρες και καταστάσεις. Ε, στο επενδυτικό σχέδιο υπάρχει ο πρώτος πυλώνας για τα χρηματοδοτικά κίνητρα και ο δεύτερος πυλώνας για τεχνική βοήθεια. Υπάρχει όμως και ένας σημαντικός τρίτος πυλώνας που αφορά το επιχειρηματικό περιβάλλον. Εάν και, τι λένε οι επενδυτές, αν μιλήσεις με αυτούς, πιστεύουν ότι τα περισσότερα εμπόδια για την επένδυση σε αναπτυσσόμενος χώρος είναι λόγω του επιχειρηματικού κλίματος και όχι λόγω το, της έλλειψης των χρηματοδοτικών κινήτρων. Δουλεύουμε από αυτού, ούτω ώστε να βελτιώσουμε τον, το επιχειρηματικό κλίμα, να έχουμε κανονισμούς πιο διαφανείς, με τη διαφθορά. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό, ούτως ώστε να μπορέσουν να προχωρήσουν αυτές οι επενδύσεις. Ε, τη μέρα της ανάπτυξης κάναμε μία ημερίδα ε, με τον κύριο Μπέργκ. Ε, ήμουνα ε, συμπρόεδρος. Ε, δεν παρατηρούμε απλώς, δεν στέλνουμε παρατηρητές στις εκλογές. Ε, δίνουμε και... στέλνουμε προσωπικό που υποστηρίζει αυτές τις χώρες, το αποσπούμε στα κοινοβούλια Είχαμε πάει στην Κένια και εγώ είχα μιλήσει με διάφορους βουλευτές. Τους εξηγούσα ότι εμείς, εγώ με το κόμμα μου, ας πούμε, πηγαίνουμε στην, στο εκλογικό κέντρο, ας πούμε, ε, τα ελέγχουμε όλα, παρατηρούμε το πώς λειτουργεί η δημοκρατία. Τους τα έλεγα αυτά και ήταν κατάπληκτοι. Πολλές ε, από τις αφρικανικές χώρες έχουν ε, περίπλοκα λογισμικά για να μετράνε ψήφους, αλλά σταματάει το πράγμα εκεί. Το θέμα είναι να πηγαίνεις εκεί να παρατηρείς πώς λειτουργεί η δημοκρατία στην πράξη, να είναι μια συνεχής προσπάθεια. Και ο ρόλος των ε, βουλευτών είναι πολύ σημαντικός και το τονίζουμε σε αυτούς. Πολύ σύντομη γιατί δεν έχουμε πολύ χρόνο. Η παρέμβαση που έγινε από βουλευτή για την ανάγκη να δούμε τους ε, SDGs σε όλες τις πολιτικές. Να υπάρξει δράση σφαιρικά, σωστό. Αυτό είναι η δυσκολία. Η δυσκολία στο UNDP είναι ότι εστιάζουμε σε, διάφο ε, σε διάφορες χώρες. Μας έχουν προσκαλέσει 170 περίπου χώρες ε, για να τις υποστηρίξουμε για την Ατζέντα 2030, όχι μόνο για το SDG 16, για όλους τους στόχους. Ε, για να φτιάξουν τα εθνικά ε, πλαίσια σχεδιασμού. Με τι μοιάζουν αυτά τα σχέδια για την Ατζέντα 2000. Ε, τι αντισταθμίσεις πρέπει να γίνουν, τι παζαρέματα, τι δούνε και λαβίν. Υπάρχει μία πλειάδα φορέων που διαβουλεύονται, χρησιμοποιούμε διάφορα εργαλεία μοντελοποίησης Εάν κάνει στοχή, α πούμε, τι επιπτώσει θα έχει στη συμμετοχή των γυναικών, στη μείωση τη φτώχεια κτλ. Αυτή είναι η πρόκληση τη ατζέντα. Και εμεί στο UNDP και άλλοι εργαζόμαστε όχι μόνο με τα κράτη-μέλη, τι εθνικέ κυβερνήσει, αλλά και με φορεί από αυτά τα κράτη, από πολλέ πολλές χώρε, 170 χώρε. Μία γρήγορη απάντηση για το ρόλο των κοινοβουλίων. Μιλήσαμε για το ρόλο των κοινοβουλίων ήδη στο να δώσουν ε, να εξασφαλίσουν συμμετοχική διακυβέρνηση το UNDP έχει συγκεκριμένο ρόλο για την ατζέντα SDG και εργάζεται για να ενισχύσει τα κοινοβούλια, να τα βοηθήσει να καταλάβουν ποιο είναι ο ρόλος τους, να καταλάβουν ε, ποιο είναι ο υποπτικός τους ρόλος, ο ελεγκτικός τους ρόλος, να καταλάβουν ποια είναι τα εργαλεία που στη διάθεσή τους, ώστε να επιτελέσουν αυτό το έργο και να εξασφαλίσουμε ότι όταν ελέγχουν προπολογισμού, πολιτικές κτλ. καταλαβαίνουν τους στόχους και την ατζέντα πιο γενικά. Η Τζούλια που ε, κάθεται πίσω στην αίθουσα ε, ξέρει πολύ καλά αυτό το πρόγραμμα. Υπάρχουν ε, οδηγία, χειρίδια κτλ. Υπάρχουν, υπάρχει και μια, ένας όγκος εμπειρίας για το πώς μπορούμε να υποστηρίξουμε τα κοινοβούλια τα οποία α, δεν είναι τόσο ισχυρά όσο τα κοινοβούλια που εκπροσωπούνται εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για να παίξουν αυτό τον ρόλο, τον ελεκτικό κτλ. πιο αποτελεσματικά. Ευχαριστούμε τους ομιλητές που ήρθαν εδώ, που μας είπαν τις απόψεις τους. Ε, είναι πάρα πολύ σημαντικός ο στόχος 16. Ε, ε, είναι μια κοινοτομία, μας τα εξηγήσατε. Ε, σας ευχαριστούμε πολύ γρήγορα για τη συμμετοχή σας. Θα περάσουμε τώρα στον επόμενο γύρο ομιλητών. Να έρθουν οι ομιλητές. Θα έρθει ο συνάδελφος να προεδρεύσει και εγώ θα πάω κάτω. Okay, thank you very much. We can start. Thank you, Linda. Ας ξεκινήσουμε. I would like to start now welcoming and short introducing briefly our second. Να σας παρουσιάσω συντομία το δεύτερο πάνελ. Πρώτα θα δώσουμε το λόγο στην κυρία Λίνα Ρότσα Μενοκάλ από το Overseas Development Institute. Μετά Συγγνώμη για τον τρόπο με τον οποίο θα προφέρω το όνομά σας η κυρία Ντεντάγιο Μπολάτζη Άντιο από την Oxfam και τέλος η κυρία Κλώε Τρίκο Οφάρελ από την ε, ΜΚΟ Safer World. Η κυρία Λίνα Ρότσα Μενοκάλ, καλώς ήρθατε στο κοινοβούλιο μας. Χαιρόμαστε που ήρθατε εδώ, θα σας ακούσουμε, θα, θα κάνετε την παρουσίασή σας. Σε αυτή τη σύντομη εισαγωγή μπορώ να σας πω ότι περιμένουμε με ανυπομονησία την παρουσίασή σας. Να ακούσουμε τη γνώμη σας. Η αίθουσα είναι δική σας. Περιμένουμε λοιπόν να ακούσουμε αυτά που έχετε να μας πείτε. Θα ήθελα να παρουσιάσετε και τον εαυτό σα. ποια είστε και τα λοιπά, ε, τι έχετε κάνει, αν μπορείτε. Um, Ευχαριστώ πολύ, χαίρομαι πολύ που βρίσκομαι εδώ. Δυστυχώς θα μιλήσω αγγλικά. Ονομάζομαι Αλίνα Ρότσα Μενοκάλ. Ε, από το Ινστιτούτο ε, Ανάπτυξης, το ODI. Και θα ήθελα να πω ότι και ως Μεξικανοί, αλλά και ως πολίτης Μεγάλης Βρετανίας, μπορεί να είμαι λίγο πιο γκρινιάρα από ό,τι συνήθως, ζητώ συγγνώμη. Με συγχωρείτε αν είμαι λιγότερο αισιόδοξη από ό,τι συνήθω. κάνω ένα βήμα πίσω σε σχέση με τα όσα ανέφερε το προηγούμενο πάνελ και θα εξετάσω ακριβώ αυτή την ιδέα των συμπεριληπτικών θεσμικών οργάνων και πολιτικών διαδικασιών. και την πρόκληση της υλοποίηση του στόχου SDG16. Όπως ε, είπαν και οι προηγούμενοι ομιλητές λοιπόν, τα συμπληρωτικά θεσμικά όργανα και οι πολιτικές διαδικασίες είναι ε, μεγίστη σημασίας για την μακροχρόνια ε, σταθερότητα, ειρήνη και ευημερία. Και όντως υπάρχουν πολλά εύρωστα στοιχεία εκεί έξω που ε, στηρίζουν ακριβώς αυτό, αυτή την υπόθεση. Θέλω να, να αναφερθώ σε δύο ευρήματα που προέκυψαν από την έρευνά μου στο θέμα των ε, θεσμών. Σε περίπτωση συγκρούσεων, βραχυπρόθεσμα, υπάρχει μια κρίσιμη οδός ε, μετάβασης και ένας τρόπος να ξεπεράσουμε τις συγκρούσεις είναι με το να έχουμε πιο συμπεριληπτικά πολιτικά συστήματα που, με συμμετοχή των ελίτ. Και είναι σημαντικό τουλάχιστον σε επίπεδο ελίτ βραχυπρόθεσμα μετά από συγκρούσεις να υπάρχει μια ελάχιστη συνεννόηση μεταξύ των ελίτ για να υπάρχει μια δυνατότητα διατήρηση της ειρήνης και σταθερότητας. Αυτό προκύπτει από τη βιβλιογραφία με πολύ καλά στοιχεία. Μπορώ να σας παραπέμψω αν θέλετε. Ένα δεύτερο έβριμα, μακροπρόθεσμα, ευρύτερα συμπεριληπτική ε, πολιτική τάξη που ε, βοηθούν στην ανάπτυξη πιο ανθεκτικών και ειρηνικών κρατών και κοινωνιών που τείνουν να έχουν και καλύτερη διακυβέρνηση, κυβέρνηση με περισσότερη δημοκρατία, νομοποίηση, ευημερία και χαμηλότερες ανισότητες. Όμως υπάρχουν πολύ καλά στοιχεία ως προς αυτό το ζήτημα της, ε, των μακροχρόνιων αναπτυξιακών προτύπων. Μάλιστα, ε, μία από τις πιο συνεκτικές ε, σχέσεις που μελετάτε είναι η διασύνθεση μεταξύ ειρήνης και δημοκρατίας και σταθερότητα και δημοκρατίας. Είναι σαφές ότι υπάρχει συσχέτιση από το 1960 και μετά μεταξύ δημοκρατίας και ανάπτυξης. Αν το εξετάσετε λοιπόν ιστορικά, δεν υπάρχει ούτε η μία ε, δημοκρατική χώρα, βέβαια ίσως αυτό αλλάξει. Μέχρι τώρα όμως δεν υπάρχει καμία δημοκρατική χώρα που να έχει πέσει ε, σε απολυταρχικό καθεστώς ε, από τη στιγμή που έχει φτάσει ένα συγκεκριμένο επίπεδο ΑΕΠ που συνέβη και με την Αργεντινή ε, τη δεκαετία του 1960. Επομένως, το ουσιώδες εδώ είναι ότι υπάρχει ένα τεράστιο χάσμα μεταξύ ε, αυτών των δύο συστημάτων που σας παρουσίασα, συμφωνία ελίτ ε, για να ξεπεραστούν οι συγκρούσει και να υπάρχει ένα ελάχιστο επίπεδο σταθερότητα. Αυτό είναι το βραχυχρόνιο και μετά μακροπρόθεσμα, πολύ πιο δύσκολο βέβαια να επιτευχθεί για το τι σημαίνει ακριβώ ε, αυτό το συμπεριληπτικό σύστημα. Αυτό μας οδηγεί στο βασικό ερώτημα πώς μπορούν τα όρια του πολιτικού συστήματος που μπορεί να είναι πολύ στενά και να επικεντρώνονται κυρίως ε, στη ελίτ, τουλάχιστον βραχυπρόθεσμα, να επεκταθούν, να ευρυνθούν ε, για να διαμορφώσουν μια ευρύτερα συμπεριληπτική πολιτική τάξη σε ό,τι αφορά και τις διαδικασίες και τα αποτελέσματα. Αυτό είναι που μας απασχολεί κυρίως σε ό,τι αφορά τον στόχο 16 αλλά και τον πρώτο στόχο ειρήνης ε, και βιωσιμότητας από, το, την ομάδα ε, την αρμόδια και έτσι είναι ένα πολύ καλό σημείο εστίασης. Όμως και εδώ θέτω αυτόν τον προβληματισμό. Αν υπάρχουν στοιχεία ότι ε, τα συμπεριληπτικά και αποτελεσματικά θεσμικά όργανα έχουν μεγάλη σημασία, δεν είναι τόσο σαφές ποια είναι αυτά τα θεσμικά όργανα που είναι ε, σημαντικά, πότε, σε ποιες περιπτώσεις και πώς μπορούμε ε, να τα διαμορφώσουμε. Επίση, δεν ξέρουμε ποια ακριβώ είναι η εικόνα, ποιο είναι ο στόχο. Θέλουμε όλοι να γίνουμε Δανία. Ε, δεν είμαστε σίγουροι πώς ε, η δημοκρατίες, οι σταθερές δημοκρατίες που θεωρούσαμε τουλάχιστον ε, σταθερές, πώς αντιμετωπίζουν αυτές τις κρίσεις. Υπάρχουν ε, λίγες συστημικές ε, γνώσεις σε ό,τι αφορά αυτές τις μεταβατικές διαδικασίες, όχι μόνο στον αναπτυσσόμενο χώρο, αλλά και στις αναπτυσσόμενες χώρες, αλλά και στις αναπτυγμένες. και αυτό δημιουργεί πολύ περισσότερα ερωτήματα από αυτά που μπορούμε να απαντήσουμε. Ένας από τους βασικούς ε, μοχλούς ε, ανάπτυξης Ποιοι είναι αυτοί λοιπόν ε, οι μοχλοί ανάπτυξης και οι διαδικασίες, πώς διαμορφώνουν τις δυνατότητες μεταρρύθμισης, αν αυτές οι μεταρρυθμίσεις είναι πάντα προοδευτικές πώς, σε ποιο βαθμό μπορούν συγκεκριμένες μορφές συμπερίληψης να ε, αντισταθμίσουν άλλες αδυναμίες εντός μιας χώρας σε ό,τι αφορά την ε, ελάφρυνση της φτώχειας αλλά και τις ανισότητες που είναι μια νέα πρόκληση που μας αποσχολεί περισσότερο πώς μπορούμε να εξετάσουμε συγκρούσεις, εντάσεις, διλήμματα και αντισταθμίσματα, τι ε, πείθει της ελίτ να ε, υιοθετήσουν ένα διαφορετικό πρότυπο συμπερίληψης είτε στη διαδικασία και στην λήψη αποφάσεων είτε στα αποτελέσματα και ποιος ωφελείται από ε, την κάθε διαδικασία. Ποια είναι η σωστή ισορροπία αν υπάρχει τέτοια. Και πώς μπορεί η πίεση από τα κάτω να αλλάξει το πολιτικό σύστημα και αν τέτοιου είδους οθήσεις από τα κάτω είναι πάντα προοδευτικές. Εξετάζουμε λοιπόν τι συμβαίνει σε αυτές τις χώρες, σε πολλές από αυτές τις χώρες που από τη σύγκρουση μεταβαίνουν σε μια πιο ανθεκτική μορφή κράτους και κοινωνίας. Αναγνωρίζουμε ότι προσπαθούν αυτές οι χώρες να ε, μεταμορφωθούν σε πολλά επίπεδα και με πολλούς θεμελιώδεις τρόπους. Ο ένας είναι από τη σύγκρουση στην ειρήνη. Όμως υπάρχουν και πολλά άλλα στοιχεία. Από ένα κλειστό σύστημα σε ένα πιο ανοιχτό που περιλαμβάνει συνήθως και μια διαδικασία εκδημοκρατισμού, εκλογές και το καθεξής, από την πολύ στενή ε, έννοια του έθνους περνάμε σε μια ευρύτερη ε, έννοια ε, της κοινότητας όπως τη φανταζόμαστε, ε, εστιάζουν περισσότερο στο ε, κοινό καλό, ε, στην αλληλεπίδραση, στο κράτος δικαίου και από τους αποκλεισμούς σε ένα πιο συμπεριληπτικό σύστημα. Υπάρχουν λοιπόν πολλές αλλαγές σε πολλά επίπεδα. Κάποιες από αυτές μπορούν να ενισχύουν η μία την άλλη. Για παράδειγμα, αν υπάρχει προσπάθεια να εστιάσουμε την προσοχή μας στο ε, δημόσιο συμφέρον και όχι μόνο ε, στα συμφέροντα συγκεκριμένων κατηγοριών ε, του πληθυσμού, αυτό μπορεί να ενισχύσει την έννοια της συμπερίληψης. Όμως γνωρίζουμε από ιστορική πείρα, γι' αυτό θα ήθελα να το θέσω, Ξέρουμε λοιπόν από ιστορική πείρα ότι αυτές οι διαφορετικές διαστάσεις ε, αλλαγής συνήθως δεν ενισχύουν η μία την άλλη. Δεν πάνε όλα καλά ταυτόχρονα. Θα ήταν πάρα πολύ καλό θεωρητικά, όμως στην πράξη δεν ξέρουμε πώς αυτά αλληλεπιδρούν μεταξύ τους και αν επιδρούν θετικά ή μπορούν ακόμα και να υπονομεύσουν αυτή τη διαδικασία. Στην ε, διαδικασία αυτής λοιπόν της μετάβασης μπορεί να υπάρχουν ε, διάφορα διλήμματα και εντάσεις που θα πρέπει να λάβουμε υπόψη. Υπό αυτή την έννοια, το θεματολόγιο χρηστής διακυβέρνησης είναι ιστορική σημασίας ε, για τον τρόπο με τον οποίο εξετάζει την αλλαγή όπω έχει σημειωθεί αλλού και στο πώ θα πρέπει να σημειώνεται στι αναπτυσσόμενε χώρε. Ξέρουμε και πάλι από παστρική πείρα ότι αυτές οι μεταβάσεις δεν είναι γραμμικές, ούτε ακολουθούν πάντα την ίδια κατεύθυνση. Είναι βαθιές πολιτικές ε, ε, διαδικασίες αλλαγής που είναι σύνθετες, ενδεχομένως και εξαιρετικά βίαιες. Υπάρχουν παραδείγματα. Για παράδειγμα, στη σύγχρονη Ρουάντα. Αυτό είναι ένα πολύ ενδιαφέρον παράδειγμα ε, τέτοιων εντάσεων. Ήταν πολύ επιτυχές το παράδειγμα της Ρουάντα υπό ορισμένε έννοιες ό,τι αφορά ε, την ανάπτυξη, την παροχή βασικών υπηρεσιών, τη μετάβαση από τη βία ε, στην ειρήνη, αλλά υπάρχουν πολύ σημαντικές αδυναμίες, ιδίως ό,τι αφορά τις πολιτικές ελευθερίες και ε, της έκφρασης γνώμης. Δεν ξέρουμε ποια είναι η σωστή οδός, όμως βλέπουμε ότι δεν ε, πάνε όλα καλά από την αρχή. Ε, εκλογές τώρα. Και αυτό τονίζει ορισμένες από τις δυνατότητες αλλά και εντάσεις που προσπαθώ να επισημάνω. Βεβαίως και οι εκλογές είναι απαραίτητη προϋπόθεση για τη λογοδοσία και την ευθύνη και νομοποίηση του πολιτικού συστήματος, όμως συνδέεται και με άλλες πρακτικές που μπορεί να μην είναι τόσο καθαρές και αθώες. μπορεί για παράδειγμα η διαφθορά να ενταθεί κατά τη διαδικασία εκδημοκράτησης. Δείτε για παράδειγμα τον αντίκτυπο των χρημάτων σε ε, εκλογικές διαδικασίες. Κάποιες φορές πρόκειται για νόμιμες πληρωμές, κάποιες ε, για παράνομες. Και αυτό συνδέεται με την ποιότητα της εκπροσώπησης. Και αυτό δεν αφορά μόνο τον αναπτυσσόμενο κόσμο. Η Λατινική Αμερική, για παράδειγμα, που το οργανωμένο έγκλημα πραγματικά έχει διεισδύσει στο πολιτικό σύστημα ε, και έχει κυριαρχήσει στη διακυβέρνηση σε κάποιους ε, τομεί, αλλά και στι ΗΠΑ υπήρξε μια πολύ ενδιαφέρουσα μελέτη στο Πανεπιστήμιο Πρίνστον που αναφέρει ότι ο ε, τις τελευταίες δύο δεκαετίες ο τρόπος ε, διακυβέρνησης δείχνει ότι η χώρα πόρο απέχει από τη δημοκρατία. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχει μεγάλη εξουσία του χρήματος. Σημαντικό είναι να το έχουμε αυτό κατά νου και πολλά προβλήματα συνδέονται με ε, τις κοντόφθαλμες πολιτικές που προκύπτουν από την αναλλαγή ε, στην εξουσία και πώς αυτό επηρεάζει την προσέγγιση μας από το δημόσιο συμφέρον ε, προς ε, τα συμφέροντα της εκλογικής μας περιφέρειας, για παράδειγμα. Η Σάρα προηγουμένως ανέφερε μία μελέτη του UMDP, μια εξαιρετική προσπάθεια να δούμε ακριβώς ε, τι ενδιαφέρει τον κόσμο. Αποκαλυπτικά τα στοιχεία, γιατί δείχνουν ότι ο κόσμος ενδιαφέρεται για την διακυβέρνηση. Είναι πολύ σημαντικό για τον κόσμο η διακυβέρνηση. Αν δείτε όμως τις απαντήσεις, βλέπουμε ότι αυτό που τους ενδιαφέρει περισσότερο είναι η αποτελεσματικότητα της διακυβέρνηση και του κράτους και λιγότερο τα πολιτικά δικαιώματα. Υπάρχει λοιπόν πραγματικό θέμα σε ό,τι αφορά τις προσδοκίες του λαού ε, για τα αποτελέσματα ε, μιας κυβέρνησης, της αποτελεσματικότητας δηλαδή, και στήριξη των δημοκρατικών αξιών ε, εν γενός. Ε, ανέκυψε το θέμα των κοινοβουλίων. Γι' αυτό είναι σημαντικό να αναφέρουμε ότι αν δούμε άλλες μελέτες όπως ε, το, το βαρόμετρο στην Αμερική, στην Ασία κτλ. Είναι απίστευτο γιατί βλέπετε ότι σε πάρα πολλές χώρες, ανεξάρτητα από τα επίπεδα τα εισοδηματικά, κάθε φορά και από όλα τα θεσμικά όργανα που αναφέρονται, δύο είναι οι θεσμοί που ε, την χάνουν χαμηλότερης εμπιστοσύνης, κοινοβούλια και πολιτικά κόμματα. Βλέπετε λοιπόν ότι υπάρχει μια πραγματική πρόκληση δημοκρατίας. Γιατί πρόκειται για τους κατεξοχήν φορείς ε, προώθησης ε, των ε, δημοκρατικών διαδικασιών και αυτοί είναι που τους εμπιστεύεται ο κόσμος λιγότερο. Υπάρχουν λοιπόν προκλήσεις, αυτό είναι σαφές. Η διεθνή κοινότητα πραγματικά καταβάλει κάθε προσπάθεια για να υποστηρίξει τα πιο συμπεριληπτικά πολιτικά συστήματα και θεσμικά όργανα ανά τον κόσμο. Όμως οφείλουμε να γνωρίσουμε ότι μέχρι πρόσφατα πολλή από τη στήριξη αυτή ως προς τη χρηστή διακυβέρνηση για παράδειγμα δεν ανταποκρίθηκε στις ε, προσδοκίες μας και αυτό συνδέεται και με τον τρόπο στήριξης ε, αλλαγής γιατί συνήθως βασίζεται σε πολύ συγκεκριμένες ιδέες για το πώς θα πρέπει να γίνει η αλλαγή και όχι τόσο σε μια πραγματική κατανόηση της αφετηρίας της κάθε χώρας. Τι είναι σκόπιμο και ρελιστικό για κάθε χώρα. Βλέπουμε ότι οι χορηγοί δωρητές συνήθως ε, επιμένουν ε, και εστιάζουν στη μορφή της στήριξής τους, ας πούμε στηρίζουν εκλογικές διαδικασίες και επιτροπές ε, καταπολέμησης διαφθοράς και όχι τόσο στην ουσία. Και έτσι αγνοούμε αυτό το βασικό στοιχείο, το κρίσιμο στοιχείο της αλληλεπίδρασης με ε, ε, τους επίσημους και ανεπίσημους φορείς. Πρέπει λοιπόν να δούμε πώς αυτή η χρηματοδότηση θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη ε, ρεαλιστικά την ε, πολιτική κατάσταση της κάθε χώρας. είναι πολύ σημαντικό. Ο κύριος Βίλ αναφέρθηκε στην ανάγκη ε, μεγαλύτερης ευελιξίας και πρέπει να είμαστε και λίγο πιο πειραματικοί και να δεχόμαστε και τον κίνδυνο να υπάρξουν ε, αδυναμίες και κίνδυνοι. Όμως ε, αυτό αφορά και τις χώρες ε, που ε, χορηγούν τέτοια χρηματοδότηση και προσπαθούν να στηρίξουν ε, τη θεσμική ε, μεταρρύθμιση. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάμε στον επόμενο μιλητή, την κυρία Αντεδάγιο. Θα μας κάνει μια παρουσίαση για τη μέτρηση της προόδου του SDG 16 στην Αφρική. Σας ευχαριστώ που ήρθατε. Πέστε μας και δύο λόγια για τον εαυτό σας, για σας. Χαίρομαι που θα συμμετάσχω στη σημερινή συζήτηση. Δουλεύω στην Oxfam, στη Δυτική Αφρική. Δουλεύουμε σε θέματα ισότητας, διακυβέρνησης και παρακολούθησής τους. Θα ήθελα να μιλήσω λιγάκι για το πώς η Αφρική μετράει την εφαρμογή των ε, στόχων της βιώσιμης ανάπτυξης, των SDG. Να ξεκινήσω με ένα ειδικό παράδειγμα. Πέρυσι σε μια προσπάθεια που έκανε η Γυρία για να καταπολεμήσει την ε, διαφθορά, ε, εκδόθηκε ένα σύλληψη για έναν ε, στρατιωτικό που κατηγορήθηκε ότι, ξόδεψε, ότι έκλεψε 89 εκατομμύρια ευρώ. Ε, ήθελε στην πραγματικότητα να δημιουργήσει, να καταρτήσει στρατιωτικούς με αυτά τα λεφτά. Ε, η αντίδραση των ανθρώπων ήταν σημαντική. Το πρόβλημα δεν ήταν ότι έκλεψε αυτός ο άνθρωπος ε, τόσα λεφτά, αλλά τους εντυπωσίασε το γεγονός ότι η κυβέρνηση τον κυνήγησε. Ε, έγινε μια επίθεση στο Δέλτα του Νίχυρα και του είπαν ε, ότι μπορεί να, πρέπει να επιστρέψει τα, τα λεφτά για να μην διωχθεί. Είναι σημαντικό σε οποιασδήποτε συζητήσεις για ειρήνη και ασφάλεια στο Δέλτα του Νίγηρα ε, να το έχουμε υπόψη αυτό. Και είπε η κυβέρνηση ότι είναι σημαντικό να γίνει κάτι τέτοιο. Ε, είναι πάρα πολύ περίπλοκο το θέμα στην Αφρική. Ε, όλοι συμφωνούμε ότι οι πρωτοβουλίες κατά της διαφθοράς είναι σημαντικό για να υλοποιηθεί ο στόχος SDG 16. η ειρήνη και η ασφάλεια όμως επίσης είναι σημαντικές και οι κάτοικοι του Νίγηρα, της, του Δέτα του Νίγηρα ε, πιστεύουν ότι είναι σημαντικό να προωθηθούν μέτρα κατά της διαφθοράς. Είναι πολύ δύσκολο να αξιολογήσουμε τα στοιχεία αυτά με δείκτες, ε, γιατί απλουστεύουμε τα στοιχεία. Ε, θα μιλήσω λιγάκι για την ανάγκη παρακολούθησης. Όλο αυτό των περίπλοκων στοιχείων. Ε, μιλάμε για την, τον Αφρικανικό Μηχανισμό Εξέτασης Ομοτήμων ε, για τη μέτρηση της διακυβέρνησης. Να σας εξηγήσω γιατί πιστεύω ότι μια τέτοια ποιοτική ε, αξιολόγηση είναι σημαντική. Είναι δύο οι λόγοι. από, πολλές από τις συζητήσεις εστιάζουν στη χρήση των δικτών, αντί για να συγκρίνουμε τις χώρες, ε, ή αντί για να εξετάσουμε το πώς υλοποιούν οι διάφορες χώρες τους ε, διάφορους στόχους. Ε, ο κίνδυνος είναι ότι έτσι υπεραπλουστεύουμε. Επίσης, πρέπει να δούμε, ε, να έχουμε υπόψη μας με τι μοιάζει η διακυβέρνηση, όπως εξήγησε και ο συνάδελφος. Χρειαζόμαστε ένα εργαλείο αυστηρό για να λάβει υπόψη του τις αποχρώσεις, όλα τα περίπλοκα στοιχεία. Μπορούμε να δούμε, ας πούμε, ότι η Νιγηρία, η Κένια σημείωσαν πρόοδο ε, γιατί κάνανε εκλογές και γιατί υπήρξε μια αναλλαγή των κομμάτων στην εξουσία. Ταυτόχρονα όμως είχαμε ε, φοβερή κοινωνική και οικονομική και εθνοτική πόλωση σε αυτές τις χώρες. Επίσης χώρες όπως η Αιθιοπία ε, έχουν κυβερνήσεις που δεν, είναι, δεν Αντιπροσωπευτικέ α πούμε και όμως ήταν ε, αποτελεσματικές για να προωθήσουν τη βιώσιμη ανάπτυξη. Επομένως υπάρχει ανάγκη να γίνει μια συζήτηση πέρα από τους δείκτες και θα ήθελα να σας ε, εξηγήσω λιγάκι αυτόν τον αφρικανικό μηχανισμό, του τι προσπαθεί να κάνει. Ο μηχανισμός αυτός αναπτύχθηκε το 2003, έγιναν πολλές συζητήσεις για τη νέα εταιρική σχέση στην Αφρική έγινε μια συζήτηση, γινόταν τότε μια συζήτηση και για τους ε, στόχους χιλιετίας. Ε, υπάρχει μια παγκόσμια και μια ε, υπηρετική διάσταση. Είναι εθελοντικό αυτό το εργαλείο, ε, είναι σημαντικό για να μετρήσεις ε, την πρόθεση της ε, διακυβέρνησης και προσπαθούν σήμερα 34 χώρες μέσα από peer learning να χρησιμοποιήσουν τον μηχανισμό αυτό. μερικές έχουν γίνει αναθεωρήσεις. Το 2014 η Αφρικανική Ένωση κατέστησε το μηχανισμό αυτό ε, που σας είπα, τον Αφρικανικό Μηχανισμό Εξέδωσης Ομοτήμων, ε, αυτόνομο θεσμικό όργανο μέσα στην Αφρικανική Ένωση. Υπάρχουν πέντε φάσεις για την ε, αναθεώρηση. Καταρχάς η χώρα κάνει μια αυτοαξιολόγηση. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό γιατί υπάρχουν φορείς από τον δημόσιο ιδιωτικό τομέα, την κοινωνία των πολιτών. εξετάζουν τη χώρα τους εξετάζουν θέματα που θεωρούν ότι επηρεάζουν τον τρόπο με τον οποίο ασκείται η διακυβέρνηση και είναι εσωτερικός μηχανισμός παρακολούθησης της διακυβέρνησης ε, και παράγει και, τρόπο, παράγει συστάσεις για το πώς θα προχωρήσει αυτή η χώρα. Είναι σημαντικό για να αισθανθεί ο καθένας ότι του ανήκει αυτή η διαδικασία, ότι είναι τμήμα της διαδικασίας. Οποιαδήποτε πρόοδος ε, για τη διακυβέρνηση περνάει μέσα από αυτό. Η δεύτερη φάση ε, αφορά μία εξωτερική αξιολόγηση ε, Η Αφρικανική Αναπτυξιακή Τράπεζα και διάφοροι άλλοι ε, έρχονται και διάφορα άλλα θεσμικά όργανα έρχονται εκεί. Η γραμματεία πούμε, του APRM, ας πούμε, η UNECA, να δώσουν τις απόψεις τους, να διευκρινίσουν τα πράγματα, να κάνουν διαβουλεύσεις γίνεται μια συζήτηση. Η τρίτη φάση είναι η σύνταξη μιας έκθεσης αναχώρα. Υπάρχουν δύο εκθέσεις, η εξωτερική έκθεση και η έκθεση που ετοιμάζει η ίδια η χώρα. Εν συνεχεία γίνεται μια παρουσίαση της, των εκθέσεων στο φόρουμ του APRM και στους αρχηγούς κρατών, κρατών, της Αφρικανικών κρατών δηλαδή, και στο τέλος Γίνεται μια δραστηριότητα ομοτήμων. Ε, η έκθεση ε, εξετάζεται μπροστά στην Αφρικανική Ένωση και οι χώρε συζητάνε τα προβλήματα τη. Ε, κάθε χώρα, όλε οι χώρε μάλλον μαζί, τα προβλήματα τη κάθε Αφρικανική χώρα. Όταν, α πούμε, έγινε η παρουσίαση για την έκθεση της Νιγηρίας. Η Νιγηρία ήθελε παρουσιαστές και από την Κένια, πούμε, για να ακούσει α, για να ακούσει και το πώς λειτουργήσε ίδια η Κένια. Το APRM έχει μία πλήρη εξαντλητική συμμετοχική φύση. Το 2005 παρουσίασε κάποιες από τις δυσκολίες ε, και προέβλεψε ότι το 2007 θα υπήρχε, θα υπήρχε εκλογική βία στην Γέννη. ας πούμε, το 2007 συνέβη κάτι τέτοιο. Ε, το 2008 είχαν γίνει επιθέσεις στην ε, Νότια Αφρική. Ε, το APRM είχε πει στην Νότια Αφρική να αντιμετωπίσει, νωρίτερα το είχε πει αυτό, χρόνια πριν, να αντιμετωπίσει κάποια προβλήματα για να αποφευχθούν αυτές οι επιθέσεις. Ε, όταν εξετάζει το APRM ε, τις επίσημες και ανεπίσημες πηγές εξουσίας, κύκλους εξουσίας και ήταν ένα καλό εργαλείο για την ανάπτυξη διαφόρων σεναρίων. Είναι χρήσιμο ε, για να τυχθούν στρατηγικέ για, την, ε, για το μετριασμό των συγκρούσεων που είναι υπέτη γιατί με αυτόν τον τρόπο εκτροχιάζονται τα SDM. Επίσης ενθαρρύνει τον ε, εθνικό διάλογο και τους εθνικούς φορείς να μιλήσουν για τα προβλήματά τους για να εξεπρεθούν λύσεις. Αν κοιτάξουμε τον SDG 16, αυτό είναι χρήσιμο, γιατί η κάθε χώρα, ας πούμε, μιλάει, κάνει μία, ας πούμε, αυτοεξέταση. Ε, και φυσικά το πώς ε, θα υλοποιηθεί ο στόχος SDG 16 εξαρτάται από το κοινωνικό-οικονομικό επίπεδο της κάθε χώρας. Λαμβάνει υπόψη η κοινωνική μορφή, ας πούμε, και η ιστορία της κάθε χώρας. Επίσης, εμείς δεν λέμε με το APRMG ε, Νιγηρία. Πρέπει να γίνει δημοκρατική χώρα, όπως η Γαλλία, ας πούμε. Λέμε, αν θέλεις να αντιμετωπίσεις τη διαφθορά, να κάποια παραδείγματα από τον κόσμο και το πώ έχει γίνει. Οι χώρες ενθαρρύνονται να κοιτάξουν πολιτικές και προγράμματα συστήματα διακυβέρνησης, τα οποία θα πρέπει να αντιγράψουν, α πούμε, και σε καμία περίπτωση δεν προσπαθούμε να του τα φορέσουμε. Και τέλος και πιο σημαντικό, το APRM έχει μια διαδικασία εγγενή παρακολούθησης ε, των κυβερνητικών στόχων. Ε, η κάθε αναθεώρηση ε, συνοδεύεται από ένα πρόγραμμα δράσης εθνικό, με λεπτομέρειες για τα προβλήματα της χώρας, πώς αντιμετωπίζονται και ποιοι κρατικοί φορείς θα τα είναι υπεύθυνοι ας και θα τα προωθήσουν. Αυτό είναι μεγάλο πλεονέκτημα. Ε, σε διαστολή με τη χρήση των ε, δικτών. Οι δείκτες λένε αυτά έκανε η κυβέρνηση, αυτά δεν έκανε κτλ. Ε, και δεν κολλάνε κατά ανάγκη όλοι οι δείκτες με τα προβλήματα που στην πραγματικότητα αντιμετωπίζει μια χώρα, ε, ανάλογα με το είδο τη κοινωνία που έχει κτλ. Θέλω να, να πω κλείνοντα ότι παρότι το εργαλείο αυτό είναι πολύ... Είναι πολλά υποσχόμενο, δεν είναι τέλειο αυτή τη στιγμή, τεχνικά έχει πολλά προβλήματα, οικονομικά δεν έχει αρκετή κάλυψη, έχει μια στατικότητα ε, στα ερωτηματολόγια, πρέπει να υπάρξει μια επικαιροποίησή τους, όμως ο μηχανισμός αυτός και άλλα τέτοια προγράμματα ποιοτικής αξιολόγησης ε, αξίζουν την προσοχή της διεθνούς κοινότητας. Πρέπει να τα δούμε από απόσταση. Να μην προσπαθούμε συνέχεια να βρούμε δείκτες για τα πάντα, γιατί ορισμένα πράγματα δεν μπορούν να μετρηθούν μέσω δικτών. Και μια και οι κυβερνήσεις έχουν ε, τόσα πολλά, μάλλον η διακυβέρνηση έχει τόσες πολλές αποχρώσεις, ε, καλό θα ήταν να έχουμε και άλλους μηχανισμούς για να κάνουμε μια πιο σοβαρή πολιτική ανάλυση. Ε, το EPRM ε δεν είναι χρήσιμο για να συγκρίνει ας πούμε, χώρες όπως μας δίνει τη δυνατότητα να το κάνουμε αυτό η χρήση δικτών, αλλά βλέπουμε πώς λειτουργούν οι κυβερνήσεις σε διαφορετικά πλαίσια, ποια στοιχεία, ποιες πλευρές της διακυβέρνησης είναι χρήσιμες για να προωθήσουμε την ανάπτυξη και μας δημιουργούν, μας ε, δίνουν γνώσεις, μας βοηθάνε στην ε, υλοποίηση του στόχου 16, αλλά και όλων των υπόλοιπων στόχων για τη βιώσιμη ανάπτυξη. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε πολύ για αυτή την εισαγωγή και περνάμε στην τελευταία, αλλά εξίσου σημαντική παρουσίαση από την ε, εκπρόσωπο της οργάνωσης Safe World που θα μας παρουσιάσει μία ακόμα ε, πτυχή και γενικότερα, ειδικότερα το πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τους, ε, στόχους, ε, τον στόχο της 16 στην πράξη και το πώς μπορεί η κοινωνία των πολιτών να εργαστεί σε ό,τι αφορά την πρόληψη των σύγκρουσεων και η Safehold στοχεύει στην προώθηση των πολιτικών και πρακτικών σε εθνικό επίπεδο που μπορούν να ενισχύσουν την ενωτική διαδικασία. Δραστηριοποιείται σε περισσότερε από 30 χώρε, σε διάφορε περιοχέ στην Ευρώπη, στην Αφρική και την Ασία. Ο λόγο σε εσά. Εάν ε, θέλουμε ε, οι δεσμεύσει που έχουμε αναλάβει σε ό,τι αφορά τι ε, ειρηνικέ δίκες και συμμετοχικέ κοινωνίε, τότε θα πρέπει να δημιουργήσουμε γνήσια ειρήνη που θα υποστηρίζεται από δικαιοσύνη και θα πρέπει να μπορούμε να διαφοροποιήσουμε αυτή την ειρήνη από την σταθερότητα η οποία δεν είναι βιώσιμη και εφαρμόζεται δια της βίας. Η ατζέντα του 2030 έχει ένα τεράστιο δυναμικό γιατί μπορεί ε, να αξιοποιηθεί από, τα, από τις χώρες και έχουν δεσμευτεί οι χώρες και τα Ηνωμένα Έθνη αλλά και διάφορες μη κυβερνητικές οργανώσεις προκειμένου να ακολουθήσουν μια 15 ετή ε, προσέγγιση με βάθος προσέγγιση. Αλλά προφανώς αυτή είναι μια πολύ αισιόδοξη προσέγγιση ε, και προφανώς θα πρέπει να εργαστούμε σκληρά ώστε να επιτύχουμε τη σωστή εφαρμογή αυτού του στόχου ε, οπότε, και στο συγγνώμη που μιλώ λίγο γρήγορα, σήμερα λοιπόν θα σας μιλήσω αργά και κατανοητά ως προς το γιατί ε, ακριβώς περιλαμβάνεται στον στόχο SDG 16, ποιες είναι οι προτεραιότητες του ε, και ποια είναι, ποιες είναι οι κύριες απειλές απέναντι στην επίτευξη αυτού του στόχου. Καταρχήν, γιατί θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση να επενδύσει σε αυτό το στόχο, όχι μόνο γιατί υπάρχουν πάρα πολλές προκλήσεις σε παγκόσμιο επίπεδο και όχι μόνο ε, το ότι η συμπερίληψη αυτής της πολιτικής αποτελεί ένα εφαλτήριο για την ε, συνεργασία με τους άλλους φορείς σε μια σειρά άλλων ζητημάτων, αλλά και επειδή ε, διαπιστώνουμε μια σειρά από νησιτικέ τάσεις. Ο αριθμός, για παράδειγμα, των ανώπλων συγκρούσεων έχει αυξηθεί από 31 το 2010 σε 50 το 2015, ενώ ο αριθμός των εκδιωγμένων έχει αυξηθεί από 37 εκατομμύρια το 96 σε 65,3 εκατομμύρια το 2015, που αντιστοιχεί δηλαδή σε μια αύξηση της τάξης του 75% σε λιγότερα από 20 χρόνια. Επίση, περισσότεροι άνθρωποι έχασαν τη ζωή του σε ένοπλε συγκρούσει το 2014 από ότι σε οποιαδήποτε άλλο ε, έτο κατά τελευταία 20 ε, έτη, ενώ το δεύτερο χειρότερο των εισαγωγικών έτο ήταν το 2015. Ε, επίσης, άλλες ανησυχητικές αποκλήσεις έχουν διαπιστωθεί ε, σε σχέση με άλλα στοιχεία του στόχου 2000, SDG 16. Για παράδειγμα, βάσει την ε, Freedom House έχουν σημειωθεί περισσότερες επιδεινώσεις από ό,τι βελτιώσει στις χώρες μεταξύ του 2005 και του 2014 ε, και τα δύο τρίτα των 180 χωρών που εξετάζονται στο πλαίσιο του δίκτυ για την ελευθερία του τύπου στον κόσμο ε, είχαν ε, χειρότερες επιδόσεις από ό,τι το προηγούμενο έτος. Εμείς λοιπόν έχουμε αναγνωρίσει πέντε τομείς στους οποίους θα πρέπει να δραστηριοποιηθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση ώστε να επιτευχθεί η εφαρμογή στην πράξη του SDG 16 αλλά και γενικότερα των SDGs. Η Ευρωπαϊκή Ένωση λοιπόν θα πρέπει να συνεχίζει να είναι υπέρμαχος του SDG 16 ε, και στο διεθνέ επίπεδο, ειδικότερα γιατί παρότι έχει συμφωνηθεί η ατζέντα του 2030, υπάρχει ακόμα δυσαρέσκεια και αντιδράσει από τα κράτη-μέλη ε, στο Νέα Υόρκιο και ακριβώ επειδή και συνεχίζεται η συζήτηση σε ό,τι αφορά την επιχειρησιακή εφαρμογή του στόχου SDG16, η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να συνεχίσει να επιδιώκει το όραμά τη για τα όσα έχει καταφέρει μέχρι τώρα. Και θα αναφερθώ σε αυτό λεπτομερέστερα στη συνέχεια. Ε, ε, επίσης, ε, θα πρέπει η υποστήριξη αυτού του στόχου να ε, λάβει χώρα και στην εθνικό επίπεδο. Αλλά εδώ θα πρέπει να έχουν πάντα κατά νου οι φορεί τη Ευρωπαϊκή Ένωση ότι η εφαρμογή λαμβάνει χώρα ε, από διαφορετικού ε, φορεί σε διαφορετικέ ε, καταστάσει και σε διαφορετικέ χρονικέ στιγμέ. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να είναι ευέλικτη η εφαρμογή τη σχετική πολιτική, θα πρέπει να αναμένουμε μέχρι για να αξιοποιήσουμε τι κατάλληλε χρονικέ συγκυρίε και θα πρέπει να τίθεται και η κατάλληλη μακροπρόθεσμη στόχη αφού έχει τέτοιο μεγάλο βάθο χρόνου ε, ο SDG 15 ετή δηλαδή βάθος χρόνου. Και αυτό με φαίνει στο δεύτερο ζήτημα ε, που θα ήθελα να θίξω, δηλαδή το πώς ε, μπορούμε να διασφαλίσουμε την επίτευξη αλλαγής στην πράξη και πώς μπορούμε να προωθήσουμε τους φορείς της αλλαγής. Η συνένεση του κονσέρνους δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι θα ε, έχει αποτέλεσμα σε πολιτικό επίπεδο αν ε, βασιστούμε στην υφιστάμενη, στο υφιστάμενο πολιτικό πλαίσιο. Δηλαδή, ενεργό υποστήριξη των φορέων που μπορούν να επιφέρουν θετική αλλαγή θα πρέπει να αποτελέσει στοιχείο του αναπτυξιακού σχεδιασμού. Ε, αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να υπάρχει ε, να αναγνωριστούν οι φορείς που έχουν ακριβώς το δυναμικό για να επιφέρουν αλλαγή ε, στις ε, κοινωνίες γιατί τα καταπιστικά καθεστώτα δεν πρόκειται να κάνουν απλές παραχωρήσεις. Η ατζέντα λοιπόν δίνει ακριβώς έναν μοχλό για την άσκηση πιέσεων σε αυτούς τους φορείς της αλλαγής και νομιμοποιεί και τους διεθνείς εταίρους για την υποστήριξη αυτών των φορέων. Ε, σε ό,τι αφορά τώρα τη συνεργασία με τους ε, ε, άλλους φορείς, η ατζέντα του 2030 αναφέρεται ειδικότερα στην ανάγκη στενής συνεργασίας μεταξύ κυβερνήσεων, πολιτιμερών φορέων και ούτω καθεξής. Και θα είναι ε, ε, όμως απαραίτητο αυτή η συνεργασία να γίνει και σε εθνικό επίπεδο. Δηλαδή οι μεγάλες μεταμορφώσεις ε, και αλλαγές δεν θα έρθουν από έναν υπουργό, από μια κυβερνητική πολιτική, θα επιτευθούν μέσω συνεργειών σε επίπεδο κράτων, κρατών και κοινωνιών και θα πρέπει να επιτευχθεί μια κατανόηση σε ό,τι αφορά την ολιστική και κοινή προσέγγιση της αλλαγής και της μεταμόρφωσης η οποία θα αποτελέσει την ε, θα δίνει τη βασική κατεύθυνση ε, για τις ε, παρεμβάσεις και η συνεργασία θα πρέπει να περιλαμβάνει και άλλους φορείς πέραν δηλαδή αυτών με τους οποίους συμφωνούμε αλλά οι οποίοι είναι πολύ σημαντικοί. Τέταρτον θα πρέπει να υπάρξει πολύ πιο συνεκτική ε, εργασία και πολιτική, ούτως ώστε να ευθυγραμμιστούν οι ε, διμερείς, πολυμερείς ε, και εθνικές πολιτικές. Καταρχής θα πρέπει να παρασχεθεί ειδική υποστήριξη σε χώρε οι οποίε βρίσκονται ή διέρχονται μια περίοδο σύραξη. Αυτό σημαίνει ότι η διμερή υποστήριξη θα πρέπει να παρέχεται με συνεχτικό τρόπο μεταξύ των κυβερνήσεων και ε, με βάθος χρόνου. Δηλαδή δεν έχει νόημα από τη μία πλευρά να ε, ε, προωθούμε τους φορείς αλλαγή σε μία χώρα ενώ ταυτόχρονα επιτρέπουμε τις εξαγωγές όπλων στις πολιτικές ελίτ των ίδιων χωρών οι οποίες ακριβώς αντίσταται σε αυτές τις αλλαγές. Επίσης η γενική η συνάφεια της ατζέντα του 2030 σε ό,τι αφορά τις διάφορες προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε και εδώ είναι απολύτως απαραίτητο αν θέλουμε να, οι υπόλοιποι να να πιστέψουν στην σημασία αυτή τη ατζέντα. Δηλαδή, ε, δεν, θα μπορούμε να, δεν θα μπορέσει η Ευρωπαϊκή Ένωση να πιέσει τι άλλε χώρε σε ό,τι αφορά την επίτευξη προόδου σε σχέση με τη διαφθορά, εάν δεν κάνει ίδια ε, το ίδιο στα δικά τη κράτη-μέλη. Επίση, θα πρέπει να αναλυφθεί αποφασιστική δράση σε ό,τι αφορά ε, τις, τους φορείς οι οποίοι προωθούν περαιτέρω τις ε, συγκρούσεις όπως για παράδειγμα οι παράνομες χρηματικές ε, ροές. Ένα ακόμα στοιχείο είναι η υποστήριξη της δημιουργίας νέων σε δεδομένων με χάρη στην ατζέντα του 2030 έχουμε πλέον τα εργαλεία για την παρακολούθηση του αν επιτυγχάνεται πρόοδο. Ε, δεν είναι τέλειοι οι δείκτε, αυτοί οι παγκόσμιοι δείκτε, αλλά θα δημιουργούν νέα ε, δεδομένα τα οποία δεν υπήρχαν μέχρι τώρα, δεν συλλέγονταν παραδοσιακά και θα επιτρέπουν τι συγκρίσει μεταξύ ε, χωρών. Για παράδειγμα, οι δείκτε σε ό,τι αφορά την ανισότητα ή τη διαφθορά θα επιτρέψουν ακριβώ τι διαδικασίε λογοδοσία των αρμοδίων και θα μπορούσαν να παίξουν ένα βασικό ρόλο όπου θα υπάρχει αμφισβήτηση τη επίτευξη αυτών των αλλαγών. Και τα κράτη-μέλη θα πρέπει να ε, ε, προβούν σε σημαντικέ επενδύσει ε, στι δυνατότητε συλλογή δεδομένων του, ειδικότερα μέσω των εθνικών στατιστικών δεδομένων συστημάτων. Η κοινωνία των πολιτών και οι πολίτες θα πρέπει ταυτόχρονα να είναι σε θέση να παρέχουν δεδομένα, ώστε να δημιουργηθούν γενικότερα οικοσυστήματα δεδομένων που θα είναι πλουραλιστικά. Ε, και επιτρέψτε μου εδώ πολύ να, να, σας αναφέρω ότι εμείς συμμετέχουμε από την πλευρά της ε, Safer World σε ε, μία πρωτοβουλία με την ονομασία SDG 16 Data Initiative, πρωτοβουλία δηλαδή για δεδομένα, η οποία προσπαθεί με τη συνεργασία 14 οργανώσεων να βελτιώσει τους τρόπους με τους οποίους μετρούμε ακριβώς την πρόοδο προς την ειρήνη, τη δικαιοσύνη και την συμμετοχή. Ε, έχοντας αναφέρει όλα αυτά, παραμένουν παρόλα αυτά μία σειρά από απειλέ σε ό,τι αφορά την επίτευξη και την εφαρμογή του στόχου ε, SDG 16 στην πράξη. Ε, Πολλέ από αυτέ τι ε, προκλήσει, τι απειλέ εντοπίζονται σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο, όχι δηλαδή στου εξωτερικού φορεί, στου οποίου δεν έχουμε μεγάλη επιρροή. Ο βασικός, το βασικό εμπόδιο που θα μπορούσε να, να βρεθεί στο, στο στη διαδικασία εφαρμογής του SDG 16 είναι εσωτερικέ εσωτερικές μας πολιτικές. Οι πρωτόγνωροι αριθμοί μεταναστών και η απειλή των τρομοκρατικών ε, επιθέσεων ε, έχουν οδηγήσει ε, στο να λάβουν αυτά τα ζητήματα ιδιαίτερη προτεραιότητα στην ατζέντα, την πολιτική ατζέντα του κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και ταυτόχρονα βέβαια η αυτή η ανασφάλεια έχει ενισχύσει τις εθνικιστικές και ξενοφοβικές φωνές στην Ευρωπαϊκή Ένωση με αποτέλεσμα αυτό βέβαια ε, να λαμβάνονται ε, ρεαλιστικές ε, βράχοι πρόθεσμες παρεμβάσεις και να δίνεται χαμηλότερη προτεραιότητα σε πιο μακροπρόθεσμες στατικές. Η πολιτική που δημοσιεύτηκε πρόσφατα παγκόσμια ε, στρατηγική για την ε, πολιτική ασφαλείας ε, αναφέρει τους, τα κύρια στοιχεία της πολιτικής ασφαλείας και αναφέρει ότι παρότι θα πρέπει να γίνουν προσπάθειες σε ό,τι αφορά την πρόληψη των συγκρούσεων και την ασφάλεια των ανθρωπίνων ζωών, ταυτόχρονα αναγνωρίζει ότι θα πρέπει να προωθείται η ειρήνη και να εξαλειφθεί η φτώχεια. Αλλά δεν θα, σε κάθε περίπτωση να ε, παραγνωρίζεται ακριβώς αυτό ο παράγοντας της εξάλληψης της και της ε, χρηστής διακυβέρνησης προκειμένου να δοθεί προτεραιότητα σε πιο πρόθυμους στόχους. Η ε, πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Ένωσης να παράσχει εξοπλισμό σε ε, τρίτες χώρες, ειδικότερα σε ό,τι αφορά εξοπλισμό που χρησιμοποιείται σε συγκρούσεις, είναι ιδιαίτερα ανησυχητικό αναφέρει η συγκεκριμένη πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Ένωσης ότι αν δεν δοθεί μια τέτοια είδους επιστήριξη ουσιαστικά δημιουργείται πρόβλημα στην επίτευξη των υπολείπων στόχων. Παρότι αναγνωρίζουμε ε, το ότι υπάρχει, ε, η αναγνώριση της Ευρωπαϊκή Ένωση ότι υπάρχει ανάγκη να ληφθεί υπόψη και να προωθηθεί το κράτος ε, δικαίου και χρηστή διακυβέρνηση, η υποστήριξη τέτοιου είδους ε, πρωτοβουλειών δημιουργεί ανησυχία. Από τη μία πλευρά η υποστήριξη τη ευημερία των ανθρώπων θα πρέπει να υποστηριχθεί γιατί αυτή οδηγεί και στην βελτίωση τη ασφάλεια με τη σειρά τη. Ε, εάν δώσουμε, αν αντιστρέψουμε αυτή τη σειρά, ουσιαστικά ε, και οι δύο αυτοί στόχοι γίνονται πιο μακρινοί. Από την άλλη πλευρά, ε, ο στόχος είναι να υπάρχει καλύτερη θεσμική δυνατότητα για περισσότερη συμμετοχή. Και παρότι αναφέρεται γενικότερα στην δημιουργία περισσότερων ικανοτήτων στου θεσμού, αναφέρεται ταυτόχρονα στο στόχο SDG 16 και ανάγκη για περισσότερη διαφάνεια. Άρα λοιπόν η παροχή εκπαίδευση ε, στι ε, κυβερνήσει οι οποίε δεν έχουν την ε, αντίστοιχη εμπειρία σε ζητήματα διαφάνεια δεν θα προωθήσει τα πράγματα. Ενδεχομένω σε κάποιε περιπτώσει να οδηγηθούμε σε λιγότερο ειρηνικέ κοινωνίε. Παρ' όλα αυτά όμως η Ευρωπαϊκή Ένωση δίνει προτεραιότητα στις ε, θεσμικές ε, ικανότητες αυτών των χωρών χωρίς να λάβει υπόψη τις ε, διαρθρωτικές αλλαγές οι οποίες θα πρέπει να λάβουν χώρα και οι οποίες τελικά προωθούν περαιτέρω την αστάθεια σε αυτές τις χώρες. Ε, παρότι έχει υπάρξει λοιπόν ιδιαίτερη έμφαση σε αυτές τις πρωτοβουλίες SPST, υπάρχει ε, μια γενικότερη προβληματική σε ό,τι αφορά και τις πιο γενικές ε, πολιτικές. Ε, για παράδειγμα, το πρόγραμμα παρακολούθησης μέσω του οποίου θα παρασχεθεί εξοπλισμός και εκπαίδευση για τις, για τις οργανώσεις όπως στην Αιθιοπία, στην Ερυθρέα και στο Σουδάν, οργανώσεις οι οποίες είναι αρμόδιες για την διαχείριση των μεταναστευτικών ρόλων είναι προβληματικό γιατί τέτοιου είδους χώρες βέβαια έχουν συστηματικά δεν έχουν επιτύχει να ανταποκριθούν στι υποχρεώσει σε ό,τι αφορά το κράτο δικαίου και τη διαφάνεια. Άρα λοιπόν η Ευρωπαϊκή Ένωση και η ανταπόκρισή τη, η απάντησή τη στην αβεβαιότητα δεν θα πρέπει ε, να αντικαταστήσει ε, τη σημασία που έχει και η προώθηση τη δημοκρατία, ε, του κράτου δικαίου, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ακριβώ σε μια τέτοια δύσκολη περίοδο είναι σημαντικό ένα φορέ όπω η Ευρωπαϊκή Ένωση να προσπαθήσει την υποστήριξη αυτών των ε, αρχών ε, σε όλε τι γωνίε του κόσμου. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό το ζητούμενο. Το ζητούμενο είναι ότι όχι μόνο δεν μπορεί να επιτευχθεί έτσι μακροπρόθεσμα πρόοδος, αλλά υπάρχει και, υπάρχουν και πολλά αποδεικτικά στοιχεία ότι οι τέτοιου είδους τοξικές εντός εισαγωγικών εταιρικές σχέσεις ε, ε, δεν οδηγούν τελικά σε αποτέλεσμα. Η γνήσια η ε, ειρήνη υποστηρίζεται από τη δικαιοσύνη, τη συμμετοχή και τις πολιτικές ελευθερίες για όλους και αυτή, αυτή η γνώση θα πρέπει να καθοδηγήσει όλες τις δράσεις από εδώ και στο εξή και ζητώ συγγνώμη από του διερμηνείς. Ευχαριστούμε πολύ όλου του ομιλητέ. Τώρα θα θέλω να δώσουμε το λόγο στα μέλη. Αλλά και στο προηγούμενο πάνελ. Δεν ξέρω αν θέλετε να συμμετάσχετε στη σημερινή συζήτηση από το κοινό. Lina? Well, just maybe to say, um, I thought it's... Περίτω να πω ότι βρισκόμαστε στην αρχή μιας διαδικασίας ε, όπου όλοι ξέρουμε πόσο σημαντικό είναι και πώς όντως πρέπει να γίνει. Ε, όμως με ενδιαφέρον βλέπουμε πώς οι δικές τους οργανώσεις όντως αξιολογούν και μετρούν ε, στην πράξη ε, τα πράγματα. Εγώ ανησυχώ η τελευταία κοινή αντίληψη για την ανάπτυξη το 2005 ε, διαμορφώθηκε σε ένα πολύ πιο ευνοϊκό και αισιόδοξο περιβάλλον. Υπήρχε ελπίδα, ε, άνοδος της δημοκρατίας σε πολλές χώρες. Όλοι είχαν την αίσθηση ότι τα πράγματα αλλάζουν προς το καλύτερο. Σήμερα δεν έχουμε πλέον ε, την ίδια αισιοδοξία. Ακούω λοιπόν τις ε, επικρίσεις για την ευρωπαϊκή στρατηγική και τους κινδύνους για την ανάπτυξη. Όμως τα πράγματα αντικατοπτρίζουν και την εκάστοτε εποχή. Και ε, σήμερα μιλούμε για την ασφάλεια, γιατί ζούμε σε έναν ιδιαίτερα ανασφαλή κόσμο. Σήμερα το πρωί είχαμε μία ακρόαση, μια κοινή συνεδρίαση με την Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων για τη Συρία. Ο Στίβεν Ομπράιαν και ο Στάφαν Τεμιστούρα μίλησαν για τα όσα συμβαίνουν αυτή τη στιγμή στη Συρία. Και πολύ ειλικρινά μπορώ να σας πω ότι χωρίς ε, ασφάλεια εκεί για τους πρόσφυγες θα, η ζωή τους τίθεται σε κίνδυνο. Έτσι έχουν τα πράγματα. Πλέον ε, υπάρχει μία ε, μεταβλητότητα που δεν υπήρχε το 2005. Επομένως, λογικό είναι να αλλάξει και η στάση μας ως προς την πολιτική και βέβαια πρέπει να μιλήσουμε για πράγματα που τα οποία δεν αρέσουν τόσο πολύ σε εμά ε, που εργαζόμαστε σε την Επιτροπή, αλλά πρέπει να έχουμε και κατά νου και τις ε, προκλήσεις και τους κινδύνους. Για παράδειγμα, υπήρχε εκείνο το έγγραφο τότε για το Αφγανιστάν που ανέφερε πολύ συγκεκριμένα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι κατανοούμε το, το θέμα, πρέπει να ασχοληθούμε με το προσφυγικό, αλλά δεν μπορούμε να δεχθούμε ε, αναπτυξιακή βοήθεια να στρέφεται προς τα εκεί. Δεν είναι αυτός ο σκοπός της αναπτυξιακής βοήθειας και των κονδυλίων. Αλλάξαμε λοιπόν τη στάση της Επιτροπής τότε. Είμαι πιο θετική, πιο ε, δεκτική στο να συζητήσουμε ε, ζητήματα ασφάλειας, αλλά θα πρέπει κάποια στιγμή να το κάνουμε. διακυβέρνηση λοιπόν θα είναι κάτι το οποίο θα μας απασχολήσει πολύ τα επόμενα χρόνια, αλλά είμαι λίγο απεσιόδοξη αυτή τη στιγμή. Συμπροεδρεύω και της ε, ομάδας ε, για τις, τους παρατηρητέ. εκλογικούς παρατηρητές. Βλέπουμε λοιπόν χώρες που στέλνουμε αντιπροσωπείες και συνέχεια έχουμε ε, τέτοια περιστατικά ανησυχητικά, όπου λέμε ακυρώθηκαν οι εκλογές ε, γιατί ο πρόεδρος αποφάσισε να κάνει τέταρτη θητεία κτλ. Υπάρχουν τέτοια ανησυχητικά φαινόμενα. Όμως ε, γνωρίζουμε ότι πρόκειται για ένα σύνθετο περιβάλλον. Ε, σημαντικό αυτό που είπατε για το Δέλτα του Νίγηρα και τα όσα είπατε ε, για το ότι πρέπει να κοιτάξουμε λίγο τα όσα συμβαίνουν εδώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση πώς γίνεται τα φορολογικά μας να, είναι τέτοιος, ε, να γίνεται τέτοιος χαμός. Να δούμε τα έγγραφα του Παναμά, ε, τους φορολογικούς μας νόμους, πριν πάμε και ε, κάνουμε συστάσεις σε άλλους για αυτά τα θέματα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Πρέπει να μείνουμε σε επαφή. Και εμένα με ενδιαφέρει η σύγκριση δεδομένων. Δεν μπορούμε να συγκρίνουμε μια χώρα σε σύγκρουση και να αξιολογήσουμε πώς υλοποιεί τους ε, στόχους βιώσιμης ανάπτυξης ε, και να τις συγκρίνουμε με άλλες χώρες που ε, τα πράγματα είναι πιο ομαλά. Μια ευρωπαϊκή χώρα, ας πούμε, με μια χώρα σε σύγκρουση. Πρέπει να συγκρίνουμε, για παράδειγμα, την Ιγυρία με την Κένια. Αυτό είναι το ενδιαφέρον. Γιατί τότε έχουμε μια εικόνα για το ποιο ε, είναι αποφασισμένο και ποιο όχι. Συγγνώμη που δεν υπήρχε μεγαλύτερη παρουσία από τους ευρωβουλευτές. Ε, δεν ε, σημαίνει αυτό τίποτα για την ποιότητα των παρουσιάσεών σας. Από την Επιτροπή, παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ. Από την Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης, αλλά συνεργάζομαι με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή εδώ και πολλά χρόνια, επομένω δεν υπάρχει πρόβλημα. Θα προσπαθήσω να είμαι σύντομο. Στην πρώτη παρουσίαση με ενδιέφερε αυτό το θέμα. Να εστιάσουμε δηλαδή όχι μόνο στις μορφές ε, δημοκρατίας και τη κυβέρνησης, αλλά και στην ουσία. Είναι πολύ σωστή παρατήρηση. Εμείς προσπαθούμε να βασιστούμε σε ορισμένες διαδικασίες που ενδέχεται να οδηγήσουν ε, στον εκδημοκρατισμό και στη χρηστή διακυβέρνηση. Είναι σημαντικό λοιπόν να υπάρχει διάλογος με τις αρχές σε πολλά επίπεδα και με τα ενδιαφέρμενα μέρη και την κοινωνία των πολιτών, πολιτικά κόμματα κτλ. Είναι πολύ σημαντικό αυτό γιατί το θέμα δεν είναι μόνο να γίνονται εκλογές, ή να θεσπίζεται μια επιτροπή κατά της διαφοράς. Ε, πολύ σημαντικό είναι το περιεχόμενο όλων αυτών και εδώ έχει ιδιαίτερη σημασία ο διάλογος. Άλλο σημαντικό εργαλείο είναι η χρηματοδοτική στήριξη. Νομίζω ότι είναι πολύ ισχυρό μέσο γιατί ενισχύει κράτη, όχι απαραίτητα εθνικά κράτη, αλλά και τοπικές αρχές να θεσπιζεται μια επιτροπη κατα τη διαφορας ε πολυ σημαντικο ειναι το περιεχομενο ολων αυτων και εδω εχει συστήματα λογοδοσίας ως προς ε, τη διαχείριση των δημοσίων οικονομικών κτλ. Όλα αυτά λοιπόν έτσι μπορούν να ελεγχθούν ως προς την υλοποίηση των στόχων και με τη λογοδοσία. Πιστεύω λοιπόν ότι δεν πρέπει να μείνουμε μόνο στους τύπους, αλλά να πούμε περισσότερο στην ουσία, στη διαδικασία που θα φέρει την αλλαγή για τους πολίτες. Το ίδιο θα μπορούσα να πω και για τον μηχανισμό αξιολόγηση ομοτήμων για την Αφρικανική Ένωση. Συμφωνώ ότι είναι πολύ ενδιαφέρουσα η διαδικασία. Γιατί γίνεται έτσι κτήμα των Αφρικανικών χωρών όλη αυτή η διαδικασία και σε όλο το κοινωνικό φάσμα. Ωστόσο, κατά πάσα παραμένει ένας βαθμός μακροχρόνιων διαδικασιών, χρονοβών διαδικασιών, και έτσι δεν λύνονται τα προβλήματα αρκετά γρήγορα. Επομένω, πρέπει να δούμε την ίδια τη διαδικασία και πώς μπορεί να ε, ενισχύσει τη συμμετοχή των φορέων. Τέλος, για την παρουσίαση της Safer World. Για τις πέντε συστάσεις που έχετε για την Ευρωπαϊκή Ένωση, νομίζω ότι μπορούμε να ε, τους προσπογράψουμε πλήρως. Αλλά Τώρα για τις επικρίσεις σας, για το πόσο αυτή η ε, σφαιρική προσέγγιση μπορεί να οδηγήσει προς διαφοροποίηση των πόρων και σε μία προσέγγιση που κατά γνώμη σας δεν είναι τόσο ελκυστική, να πω ότι πρώτα απ' όλα για αυτή την στρατηγική. Το 2003 υπήρχε μία ασφάλι... στρατηγική ασφάλεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τώρα έχουμε ε, σφαιρική στρατηγική για την ε, άμυνα, την ασφάλεια και αυτό δεν συνδέεται μόνο με τον ε, τίτλο, είναι και θέμα ουσίας, αλλά αφορά και τη βιώσιμη ανάπτυξη σε όλο τον κόσμο. Ε, προώθηση και ενίσχυση της ανθεκτικότητας για να έχουμε θετικές αντιδράσεις από χώρες που είναι κοντά μας, γύρω μας, στα σύνορά μας. Μετά, σε ό,τι αφορά τη μετανάστευση για την ασφάλεια. Με ορισμένε χώρες έχουμε ξεκινήσει εταιρικέ σχέσεις πλαίσια. Υπήρχε μια σημαντική όθηση να έχουμε αποτελέσματα σε ό,τι αφορά τις ε, συμφωνίες ε, επιστροφής και επανεισδοχής με αυτές τις ε, χώρες. Όμως, βλέπουμε ότι διαμορφώνεται και ένας αμφίδρομος διάλογος δεν είναι μόνο ότι ενισχύουμε συγκεκριμένε μορφέ δραστηριοτήτων, βραχυπρόθεσμα, μακροπρόθεσμα. Όχι, αλλά, ε, και σε κάποιες από αυτές τις ε, χώρες εταίρους ε, βλέπουν, ε, βλέπουμε και σε εκείνους κάποιο όφελος. Αν στις χώρες του Σαχέλ βλέπουν λοιπόν ότι μπορούμε να τους βοηθήσουμε σε ό,τι αφορά τη διαχείριση των συνόρων τους, και εκείνοι λοιπόν θεωρούν σημαντικό για τη σταθερότητα της χώρας τους για την επιμερία, για παράδειγμα, ε, των ε, πολιτών στις ακριτικές τους περιοχές. Ζητούν λοιπόν από την Ευρωπαϊκή Ένωση να τις ε, στηρίξει για την καλύτερη διαχείριση των συνόρων, ε, να στηρίξει τις ε, τοπικές αρχές, τις περιοχές αυτές όπου δεν υπάρχει τόσο έντονη παρουσία του κράτους. Θα έλεγα λοιπόν ότι το θέμα δεν είναι τόσο να επιβάλλουμε στόχους και θεματολόγια, αλλά να συμμετάσχουμε κι εμείς ε, στην υλοποίηση ενός θεματολογίου που μπορεί να είναι δύσκολο να υλοποιηθεί για την κοινή γνώμη και στις χώρες μας και σε εκείνες τις χώρες, αλλά που συμπεριλαμβάνει στοιχεία μη υποφελή και για τις δύο πλευρές. Αντίστοιχα και σε ό,τι αφορά την στήριξη ε, ικανοτήτων για τους ε, φορείς ασφαλείας ε, σε πολλές από αυτές τις χώρες, αναπτυσσόμενες ή όχι, αυτοί, αυτές οι δυνάμεις ασφαλείας μπορούν να αποτελέσουν από τη μία απάντηση στην αστάθεια, από την άλλη μπορούν να βρίσκονται και στην αιτία της αστάθειας. λόγω διαφθορά και το καθεξής. Επομένω, το να στηρίξουμε τις μεταρρυθμίσεις ε, στον τομέα τη ασφάλειας, της διαφάνειας, της λογοδοσίας σε αυτούς τους θεσμούς, είναι κάτι που βοηθάει όχι μόνο τις ίδιες τις δυνάμεις ασφαλείας, αλλά γενικότερα τη σταθερότητα, τη λογοδοσία, ενδεχομένω και την ειρήνη σε κάθε χώρα. Γνωρίζετε, πιστεύω, τις ε, πολύ συγκεκριμένες ε, καταστάσεις ε, και τις προϋποθέσεις που θέτουμε εμείς. Δεν είναι μια γενικόλογη στήριξη για τις δυνάμεις ασφαλείας. Όμως μιλούμε, λέμε ότι θα πρέπει να εντάσσεται σε ένα ευρύτερο πλαίσιο και πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων, με εποπτεία, με λογοδοσία σε ό,τι αφορά τη διαχείριση. Και εδώ λοιπόν υπάρχει δυνατότητα μιας ε, αμοιβαία υποφελούς διαδικασίας όπου παρέχουμε στήριξη που θα ε, συμβάλλει στην ε, σταθεροποίηση, την ασφάλεια και στη λογοδοσία. Και αυτό μπορεί να γίνει και σε τη φορά τα ζητήματα ο ε, και ΝΤΑΚ κτλ. Ευχαριστώ για τις παρατηρήσεις. Ο κύριος Ολιβιέ από τη Γενική Διεύθυνση ΔΕΒΚΟ. Πολύ σύντομα να συμπληρώσω της, ε, την παρέμβαση του συναδέλφου της ΙΕΣ. Υπάρχει μια ανακοίνωση που ανέφερε ο συνάδελφος στην παρουσίασή του, που κανένας άλλος δεν ανέφερε, σας ευχαριστώ την προσοχή σε αυτή την ανακοίνηση. Και στα σχετικά συμπεράσματα του Συμβουλίου. Είναι η βάση για την ασφάλεια των ανθρώπων μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα ανάλογα με το πλαίσιο της κάθε χώρας, με αίσθηση ότι σου ανήκουν αυτά τα πράγματα, ότι συμμετέχεις στην διαμορφωσή τους και με αρχές δημοκρατικής διακυβέρνησης. Είναι το μεταπλαίσιο της υποστήριξής μας και το έχουν επικυρώσει όλα τα κράτη-μέλη και πρέπει να το υπενθυμίσουμε. Συμμετείχα στην ομάδα που το συζήτησε και προσπαθήσαμε να απεμπλακούμε από συγκεκριμένα πλαίσια, παρότι δεν είναι εύκολο να προσπίσει ότι δεν υπάρχουν συγκεκριμένα πλαίσια και ότι συζητάσαν κενό. Η πρωτοβουλία CBS εντάσσεται σε αυτό το πλαίσιο. Να υπενθυμίσω μια και συνεχίζεται η συζήτηση και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα πρέπει να συζητήσει το CBS2. Ε, το έχουμε υπόψη, είμαστε στη μέση της συζήτησης και θα γίνει αυτή η συζήτηση. Ευχαριστούμε. Κοιτάω και το χρόνο. Θα δώσω δύο, δύο μισή σε κάθε μία από τις ομιλήτριες για να απαντήσουν. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ για τις ερωτήσεις και τα σχόλιά σας. Πολύ σύντομα να απαντήσω σε όλους. Με ένα σχόλιο. Φυσικά συμφωνούμε ότι είμαστε σε διαφορετικό πλαίσιο και είναι πολύ σημαντικό να συγκρίνεις το, την Ευρωπαϊκή Στρατηγική του 2000, για την ασφάλεια του 2013 με την Παγκόσμια Στρατηγική που μόλις υιοθετήθηκε. Ε, είναι τελείως διαφορετικά τα πλαίσια και αν θυμάμαι καλά, στο 2013 λέγανε ότι ποτέ δεν ήταν τόσο ευημερούσα, τόσο ειρηνική η, ευημερ... η Ευρωπαϊκή Ένωση και τώρα τρία χρόνια μετά το 2016 είμαστε σε υπαξιακή κρίση. Το πλαίσιο είναι τελείως διαφορετικό, αναγνωρίζουμε ότι πρέπει να σκεφτούμε διαφορετικά λοιπόν. Και νομίζω ότι έχουμε και την ευκαιρία να δουλέψουμε καλύτερα, να είμαστε πιο αποτελεσματικοί σε αυτά τα πολύ περίπλοκα θέματα. Εγώ διάβασα πολλές από αυτές τις ευρωπαϊκές στρατηγικές, πέρασμα του Συμβουλίου, ανακοινώσεις ε, χαίρομαι που τις διαβάζω, γιατί έχουν όλα τα βασικά συστατικά που ζητάμε εδώ και χρόνια. Ε, ανθρώπινη ασφάλεια, ε, ευαισθησία απέναντι στο φύλλο και χαίρομαι που ε, δουλεύουμε σε ένα περιβάλλον όπου οι άνθρωποι για τους οποίους κάνουμε λόμπι καταλαβαίνουν τι εννοούμε εμείς και τι λέμε. Θέλω όμως να είμαστε σίγουροι ότι αυτές οι αρχές ε, εμπλέκουν την Ευρωπαϊκή Ένωση το συνόλο της. Και σε διπλωματικό επίπεδο, αλλά και σε τοπικό επίπεδο προγραμμάτων, ας πούμε. Ε, συνεργαζόμαστε με την ΤΕΦΚΟ για κάποιες κατευθυντήριες γραμμές για τη σημασία που έχει το είδος της σύγκρουσης. Στο μέλλον τα προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ελπίζω να, να λαμβάνουν περισσότερο υπόψη ε, το είδος της σύγκρουσης ε, και πώς οι παρεμβάσεις μπορεί να έχουν αρνητική επίπτωση είτε άμεσα είτε αργότερα. Δεν έχει νόημα να λαμβάνουμε υπόψη το είδο τη σύγκρουση μόνο σε διπλωματικό επίπεδο. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ε, και η διεθνή κοινότητα προσπαθεί να δημιουργήσει ε, υποδομέ κράτου και ανθεκτικότητα στο Σουδάν. Παράλληλα, πρέπει να ενισχύσουμε το δυναμικό τη χώρα για να αντιμετωπίσει, για να διαχειριστεί τα σύνορά της. Μην ξεχνάμε όμω ότι αυτή είναι η χώρα που έδιωξε άλλου από το εσωτερικό της πρέπει να δείξουμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση σέβεται τις αρχές, σέβεται την ανθρώπινη ασφάλεια, γιατί τελικά ελπίζω να παρεμβαίνουμε στο Σουδάν, ούτω ώστε οι Σουδανέζοι να ζήσουν πιο ειρηνικές φορές. Και δεν λέω ότι το να έρθουμε σε, σε επαφή με τους Σουδανέζους και τα λοιπά δεν θα έχει θετικά αποτελέσματα και καλά, απλώς λέω ότι είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί. Um, ευχαριστώ για τα σχόλιά σας. Συμφωνώ ότι το IPRM είναι πολύ χρονοβόρο. Για τον πρώτο στόχο είναι σημαντικό όμως. Είναι σημαντικό να πάρουμε το χρόνο και να διατρέξουμε την πρόσφατη ιστορία της κάθε χώρας, κάποια από τα θέματα που, και προβλήματα που αντιμετωπίζει είναι προϋπόθεση ούτω ώστε να αποκτήσουμε μια καλή ιδέα για την περιπλοκότητα ε, που, και το πλαίσιο της κάθε χώρας. Ε, μετά από αυτές τις α, εκτεταμένες αναθεωρήσεις, ας πούμε, ε, όπως Κένια, πούμε, πέρασε από μια τέτοια εκτεταμένη αναθεώρηση, μετά μπορούμε να περάσουμε σε πιο ευσύνοπτες αναθεωρήσεις, ε, για να βλέπουμε πώς σημειώνεται πρόοδο για τα διάφορα θέματα που αναφέρει το APRM. Καταρχάς, ε, έχει σημασία και η ποσότητα των αναθεωρήσεων και η ποιότητα. Μπορούμε να χρησιμοποιούμε εναλλάξ, ας πούμε, κάποιες πιο ενδελεχείς ε, αναθεωρήσεις, επισκοπήσεις κλπ. και κάποιες πιο συνοπτικές. Οι αφρικανικές χώρες είναι αρκετά διαφορετικές. Άλλο η Σενεγάλη, άλλο η ακτή του Ελεφαντοστού, άλλο η Κένια. Όλες έχουν μεταπικιοκρατική ιστορία, αλλά έχουν διαφορετικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν. Ε, η σημασία του APRM είναι ότι οι Αφρικανοί μιλάνε μεταξύ τους. Έχει σημασία να, να ακούσουμε τι λένε οι ίδιοι Αφρικανοί για την καλή διακυβέρνηση στις χώρες τους. Ενθαρρύνουμε χώρες να δουν τρόπους, να βρουν τρόπους για να αντιμετωπίσουν τα προβλήματά τους και στην Αφρική και αλλού. Δεν ζητάνε από του Αφρικανού να εστερνιστούν μια φιλοσοφία για την καλή διακυβέρνηση, αλλά να αναπτύξουν μια φιλοσοφία για το τι είναι η καλή διακυβέρνηση. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Η διακυβέρνηση δεν είναι, δεν είναι μια μαθηματική εξίσωση, υπάρχουν αμφισβητήσει. Ο Νότο τη Σενεγάλη, α πούμε, δεν θεωρεί δεν βλέπει τη διακυβέρνηση, ας πούμε, με τον ίδιο τρόπο όπως η Βόρεια Σενεγάλη. Υπάρχουν πάρα πολλέ ευαισθησίε και στο εσωτερικό μια χώρα και όλα αυτά πρέπει να τα λάβουμε υπόψη μα. Ευχαριστώ όλου. Η δεκαετία του 90 ήταν ε, μια δεκαετία αισιοδοξία. Είχα τελειώσει, είχαμε φτάσει στο τέλο τη ιστορία. Ε, είχαμε φτάσει στη δημοκρατία. Το 2005 ήμασταν λιγότερο αισιόδοξοι. Είχαμε ήδη δεχτεί τις τρομοκρατικές επιθέσεις στις ΗΠΑ, και ο πειραματισμός με τον εκδημοκρατισμό δεν είχε προχωρήσει όπως περιμέναμε. Και τώρα φτάσαμε στο τέλος του οράματος. Ζητώ συγγνώμη που είμαι τόσο απεσιόδοξη. Αλλά τι να σας πω, δεν μπορώ να σκεφτώ τίποτα άλλο. Μετά το Brexit πραγματικά ε, έχω πέσει σε ζωφερά πελάγη απεσιοδοξίας. Φτάσαμε σε μια στιγμή κρίσιμη, μια στιγμή που όπου αμφισβητούν τα πάντα για το πώς θα προχωρήσουμε. Και στο Ηνωμένο Βασίλειο και στι Ηνωμένε Πολιτείες είδαμε μία δυσαρέσκεια τη δυσαρέσκεια των ανθρώπων α, όταν περιμένουν κάποια πράγματα από τις δημοκρατίες και οι δημοκρατίες αυτές δεν τα υλοποιούν. Και όλα αυτά στα οποία πιστεύαμε και στην Ευρώπη και στην Αμερική, πράγματι δεν είναι τόσο ιερά και παραβίαστα πια. Ε, είναι σημαντικό αυτό να το δούμε και το μέλλον. Ε, είναι σημαντικό και για την ποιότητα της ε, εκπροσώπησης, δημοκρατικής ή όχι. Ένα από τα πράγματα που μου κάνει εντύπωση είναι το Ίδρυμα Μπέρκοφ, που είναι ένα γερμανικό ίδρυμα που έκανε μια πολύ καλή δουλειά για λογαριασμό του ΟΣΑ. Για το πώς οι δωρητές ε, προώθησαν τον στόχο 1 για τη δημιουργία θεσμικών οργάτων ε, χωρίς αποκλεισμούς. Το μήνυμα που δίνεται είναι κάτι ότι δεν υπάρχει τίποτα το καινούριο, ε, τίποτα το καινοτόμο. Έχουμε τα ίδια, τα ίδια που έχουμε δει και ξαναδεί και τα λοιπά, ποσοστώσεις. πρέπει οι πολιτικές διαδικασίες να χτιστούν πάνω σε διάλογο. Είναι σημαντικό αυτό. Έτσι πρέπει να προχωρήσουμε. Και οι δωρητές, η Ευρωπαϊκή Ένωση, η UNDP και άλλοι μπορεί να χρησιμοποιήσουν την επιρροή τους ε, όχι μόνο για να δίνουν χρήματα, αλλά για να παρέχουν ένα χώρο όπου θα αναπνέουν οι εσωτερικοί φορείς, θα μπορούν να συζητάνε κτλ. Για να μπορέσουν από κοινού συλλογικά να ξεπεράσουν διάφορα προβλήματα. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Um, να πω και ένα θετικό. Δεν ξέρω αν ξέρετε τη Γουατεμάλα, αν ξέρετε τι έχει συμβεί. Υπάρχει ένα φρικτό στρατιωτικό αυταρχικό καθεστώς. Μετά από αυτό δημιουργήθηκε μια διαδικασία πάρα πολύ ευχάριστη, αισιόδοξη, οικοδόμησης ε, της ειρήνης. Τριάντα χρόνια μετά έγιναν κάποια, κάποιες θεμελιακές αλλαγές. Μετά από κάποια σκάνδαλα διαφθοράς που ξέσπασαν ας πούμε, ε, χάρη στην καλή και πολύ συνετή παρέμβαση του ΟΗΕ και μοναδική μάλιστα, πουθενά άλλου δεν έχει δοκιμαστεί, πουθενά άλλου δεν έχει γίνει, ε, χάρη σε μία προσέγγιση bottom-up και top-down ε, μπορέσαμε να αντιμετωπίσουμε κάποιες από τις ε, ρίζες του προβλήματος. Ίσως σε 10 χρόνια σας πω άλλα, αλλά εν πάση περιπτώσει το θετικό. Γιατί τη Γουατεμάλα. Κάποιες ε, διαδικασίες ε, αλληλεπίδρασης, διαλόγου κτλ. είναι πολύ σημαντικές και καλό πράγμα είναι η Γουατεμάλα. Ευχαριστώ. Κλείνουμε εδώ. Ήταν χρήσιμο όλα αυτά πολύ για τη δουλειά μας. Ε, για την Ευρωπαϊκή Συνένωση για την Ανάπτυξη, ε, για το πλαίσιο μετά το Κοτονού κτλ. Ναι, υπό το σημείο 14 δεν έχουμε κάποιες ερωτήσεις, οπότε δεν χρειάζεται κάτι άλλο υπό τα διάφορα. Ε, να αξιοποιήσω την ευκαιρία και να ευχαριστήσω δύο μέλη που είναι η τελευταία του συμμετοχή γιατί έβγε από την ε, σοσιαλιστική ομάδα και συνεργαστεί με όλους τους συναδέλφους εδώ και με την γραμματεία και έχει κάνει ε, πολύ καλή δουλειά στο αναπτυξιακό τομέα ε, οπότε θα εργαστεί τώρα στην ΤΕΦΚΟ οπότε αυτό που χάνουμε εμείς με την απουσία του το κερδίζετε εσείς με την παρουσία του και δεύτερον ο Τρίσταν Στόψμα χρειάστηκε να αποχωρήσει από την αίθουσα, αλλά και γι' αυτό ήταν η τελευταία ε, συνεδρίαση. Είναι από τα θύματα, αν θέλετε, του Brexit. Ε, θα επαστρέψει λοιπόν ε, στο Ηνωμένο Βασίλειο και είναι κρίμα γιατί πραγματικά έκανε εξαιρετική δουλειά εδώ και αποφεληθήκαμε από την εμπειρία του. Είναι ευλογητό ότι χάνουμε αυτού του δύο συναδέλφου. οι δύο επόμενε συνεδριάσει, καταρχήν κοινή συνεδρίαση, δεν έχουμε επίσημη δική μα συνεδρίαση μέχρι τον Ιανουάριο. Το, την Δευτέρα λοιπόν στι τρει κοινή συνεδρίαση με την ΑΦΕΤ σε ό,τι αφορά την περιοχή των μεγάλων λιμνών στην Αφρική. Και εδώ τα πράγματα δεν είναι πολύ θετικά, μάλλον τη να είναι. Ε, και στις μισή θα έχουμε μία ε, συζήτηση εκεί με τους με τους ε, λευκόκρανους από την Κένια και θα έχουμε και την περαιτέρω ενημέρωση σε ό,τι αφορά και τη Μοσούλη και την Αλέπο. Έχουμε λοιπόν ε, από εκεί και μετά την κοινή συνάντηση με ΑΦΕΤ και Ντρουά σε ό,τι αφορά το γραφείο ε, Ζαχάροφ ε, και την, το γεγονό ότι απονεμήθηκε στις γυναίκες ζήτη που είχαν τύχει διαφορών κακοποιήσουν από το Ισλαμικό κράτος επόμενη συνεδρία στις 26 Ιανουαρίου και ευχαριστώ και τους Γερμανείς για τα 5 συμπληρωματικά λεπτά που μας έδωσαν. Έτσι καλώς δεν θα μας δείτε το δικαιωμένο οπότε σας ευχαριστώ όλους και ευχαριστώ όλους τους ομιλητές εδώ του πάνελ.